Bom dia a todas e a todos. Vamos começar a nossa reunião, que tem hoje muitos pontos na ordem de trabalhos, incluindo nos votos. Θα αρχίσουμε με τα σημεία της ημερήσιας διάταξης. Θα αρχίσουμε με ένα πρώτο σημείο σχετικά με τον εξυγχρονισμό ε, των πολιτικών των δημοσίων συμβάσεων. Ο εισηγητής για είναι η κυρία Τζούλη Έχουμε μια εισήγηση από την Επιτροπή ΙΜΚΟ, η κυρία Ρούλε. η κυρία Τζούλι Γκίρλινγκ θα μας παρουσιάσει την έκθεση για γνωμοδότηση. Έχετε το λόγο, κυρία. Thank you, Madam um, Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους σας. Το πρώτο πράγμα είναι, δεν ξέρω, αν κάποιος από σας ε, διάβασε την πράσινη βίβλο, Όπως γίνεται με αυτές τις νομοδοτήσεις, ε, πρέπει να δούμε την χρησιμότητα της απασχόλησης μέσα στην έκθεση ε, και τι γίνεται στο, ε, με το θέμα των δημοσίων συμβάσεων. Αν μου το επιτρέπετε λοιπόν, θα δω ε, ποια, ποιος είναι ο συλλογισμός που κρύβεται από πίσω. Είναι σημαντικό να δούμε ότι ε, στην πράσινη βίβλο πρέπει να αυξηθεί η αποδοτικότητα των ε, δαπανών και είναι κάτι το που πρέπει να λάβουμε υπόψη σε αυτή την Επιτροπή είναι ότι οι διασυνοριακές δημόσιες συμβάσεις που διευκολύνονται από κανονισμούς βρίσκονται πολύ ε, πιο πίσω από τις ε, ιδιωτικέ διασυνοριακές δραστηριότητες και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει ε, να εξετάσουμε και να καταλάβουμε τους λόγους αυτής της υστέρησης. όσο αφορά την ουσία, το περιεχόμενο, αναγνωρίζω την σημασία της ε, GPA πρόκειται για την ε, συμφωνία ε, του ΠΟΕ που είναι η μόνη δεσμευτική συμφωνία που ασχολείται με τις δημόσιες συμβάσεις. Είναι, αν θέλετε, ένα έγγραφο το οποίο προσφέρει κάποιο προσανατολισμό. Πρόκειται για ένα πολυμερές έγγραφο που διέπεται από, από ένα, μια επιτροπή από μέλη του ΠΟΕ μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε λοιπόν το καθήκον και την υποχρέωση να βεβαιωθούμε ότι την χάνουν σεβασμού οι διατάξεις. Ε, υπάρχει η αρχή ότι οι διάφοροι, τα διάφορα μέρη έχουν σημαντικό ρόλο να παίξουν στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών για την καινοτομία και την βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης. Και νομίζω ότι το πραγματικό θέμα um, όχι υψηλής αξίας ευκαιρίες απασχόλησης. Όχι όμως εις βάρος των δημοσίων συμβάσεων που θα είναι λιγότερο ανταγωνιστικές και λιγότερο αποτελεσματικές για τα χρήματα που θα δαπανώνται. Είναι δυσχερές αυτό να επιτευχθεί. Ξέρω ότι ήταν δύσκολο να μπορέσει να επιτευχθεί η σωστή ισορροπία. Προχωρώντας παρακάτω, τι είναι αυτό που θεωρούμε λοιπόν ότι είναι κοινωνικό όφελος ή κοινωνικά θετικό υπό την πιο απλή έννοια και προσδιορισμό. Να δίνουμε ευκαιρίες σε αυτούς τους ανθρώπους, να διασφαλίζουμε ότι άνθρωποι όλων των στρωμα... διαστρωμα... της διαστρωμάτωσης της κοινωνικής θα έχουν ευκαιρίες. Δεν θα είναι αρνητική μεταχείριση των νέων ή των ατόμων με μειονεξίες ή ειδικέ ανάγκες ή οποιονδήποτε άλλων. Η των ατομων με μειονεξιες η ειδικε αναγκες η οποιονδηποτε αλλον η δικη μου άποψη και σκέψη είναι, είναι ότι ενώ μπορώ να υποστηρίξω πλήρως αυτόν τον στόχο πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Να μην υπάρξει κάποια, κάποιος εφησυχασμός όσον αφορά την προσέγγιση μας για αυτά τα θέματα. Έχουμε τόσα πολλά συντάξει για τις απαιτήσει για τις δημόσιες προμήθειες και αγορές που πιστεύει το κοινό ότι είναι τομέας αποκλειστικά του δημοσίου αυτός. Και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι αρχές που θα θεσπιστούν θα μπορούν να υλοποιούνται, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα. Να είναι δηλαδή για όλους οικουμενικά προσπελάσιμες αυτές οι αξίες, αυτές οι ευκαιρίες και δυνατότητες. Επίσης συνέταξα στο εδάφιο 4. Ένα άλλο σημαντικό σημείο είναι αυτό, να διασφαλίσουμε ότι οι δεξιότητες και οι απαιτήσει για την κατάτηση θα είναι Ξέρω ότι αποτελεί μέλημα της ε, ανύψωσης, αναβάθμισης των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού στην Ευρώπη, να αναγνωρίσουμε τη σημασία της δεξιότητας και να δούμε ότι αυτό πρέπει να ενδυναμωθεί, να προαχθεί. Επίσης σημειώνω ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πράγματι στην οικονομία μας ε, και τόσες φορές ε, αναφέρεται αυτό και λέμε ότι είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Εδώ πρέπει να δραχθούμε τις ευκαιρίες, να δοθεί σωστή σημασία, η σπουδαιότητα που δει σε αυτές τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για τις ε, διαδικασίες για τις ε, αγορές και προμήθειες πρέπει να απλουστευτούν οι κανόνες και οι διατάξεις. Σαφώς αυτό δεν είναι το κύριο σώμα όσον αφορά την απασχόληση σε σχέση με την έκθεσή μας. Σκέφτηκα όμως θα έπρεπε να αναφέρουμε αυτό το σημείο στην άλλη Κοινοβουλευτική Επίτροπη, διότι αυτό που δεν θέλουμε είναι να δημιουργηθεί ένα πιο περίπλοκο, πιο σύνθετο πλαίσιο. Θέλουμε κάτι πιο απλό, πιο εύκολο να το διαχειριστούμε και να προαχθεί. Θα έλεγα λοιπόν τούτων λεχθέντων αυτή είναι η κύρια, η κύριη προσανατολισμή της έκθεσής μου. Είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω ερωτήσεις. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Τζόλι Γκέλιν. Και έχουν ζητήσει δύο να παρέμβουν, η κυρία Τερμαν και ο κύριος Κοφεράτη. Η κυρία Τέρναν έχει τον λόγο, παρακαλώ. Okay, Ευχαριστώ για αυτή την έκθεση. Είναι ένα καλό σημείο αφετηρίας για μια γνωμοδότηση για θέματα απασχόλησης. Στην ΙΝΚΟ ένας πράσινος συνάδελφος έχει αναλάβει αυτό, Χάιντερ Ρούλε. Είμαι ικανοποιημένη με το έργο που έχει κάνει ήδη. Έχουμε όμως έργο ως Επιτροπή Απασχόλησης, όπως ήδη προαναφέρατε, να επικεντρωθούμε στις πτυχές της απασχόλησης ε, των ε, δημόσιων αγορών και προμηθειών. Ένα μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ, ένα μεγάλος μοχλός που αν χρησιμοποιηθεί σωστά, μπορούμε να πούμε και να τονίσουμε τι είναι η κοινωνική διάσταση σε αυτές τις διεργασίες και πώς μπορεί να επιτευχθεί. Θα ήθελα αυτά να τονίσουμε και ίσως να ε, αναπτυχθεί κάπως το σημείο των κοινωνική της κοινωνικής διάστασης. Όταν πρόκειται για αγαθά, σίγουρα έχουμε και την εμπλοκή της παραγωγής και τη συνιστόσα της ε, ζήτησης, δηλαδή η ισότιμο δίκαιο εμπόριο θα μπορούσε να πει κανεί. Για τις υπηρεσίες, όταν έρχεται ώρα να εξετάσουμε τις υπηρεσίες, υπάρχει νομική αβεβαιότητα σε σχέση με τις διατάξεις ή απαιτήσει ε, για τις ε, κοινωνικές, ε, τις κοινωνικές συνιστώσεις όσον αφορά τους όρους εργασίας και το καθήκον να εκπαιδεύουμε και να κατατίζουμε. Υπήρχαν τριβές στη χώρα μου και ίσως και σε άλλες χώρες επίσης. Τι είναι δυνατόν να γίνεται. <clears throat> Δεν θα πρέπει να στρεβλώνεται ο ανταγωνισμός. Να ζητείτε από μια εταιρεία για παράδειγμα να κατατίζει νέους μέσα στις ε, ε, δράσεις της. Όλες αυτές οι περιπτώσεις δημιουργούν μια κατάσταση όπου δεν τολμούν πλέον οι τοπικές αρχές να υπομισθούν αυτή την πτυχή της κοινωνικής ε, διάστασης στις ε, προμήθειες και αγορές και αυτό δεν είναι καλό. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα επανορθωθεί αυτό, θα αντισταθμιστεί. Θα ήθελα να προσθέσω επίσης ότι Αυτές οι αγορές είναι μία μέθοδος να στοχεύσουμε ειδικέ ομάδες, να στοχοθετήσουμε που βρίσκονται πιο απομακρυσμένες από την αγορά εργασίας, άτομα με μειονεξίες ή ειδικέ ανάγκες, μακρόχρονα άνεργοι, όλα αυτά να μπορέσουν να ενταχθούν, σε να προαχθούν σε ένα κοινό πλαίσιο. Ως Επιτροπή απασχόληση ίσως θα έπρεπε να κάνουμε ένα σύντομο σχόλιο για τις ε, ταξινομήσεις ε, B και να, τους λόγους για τη διατήρηση αυτής της ταξινόμησης. Επίσης, όσον αφορά τις, α, τη σύγχυση που δημιουργείται σε σχέση με τους κανόνες και τις διατάξεις πρέπει να αντιμετωπιστεί και αυτό το πρόβλημα. Τελευταίο σημείο, να αναφερθούμε στην καινοτομία επίσης, διότι έχει σημασία κλειδιού για την δημιουργία θέσεων απασχόλησης μπορεί να βοηθήσει να υλοποιηθούν κύριοι στόχοι για την απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για την απασχόληση αλλά για την καινοτομία επίσης. Μπορούμε να δημιουργήσουμε αυτή τη διασύνδεση, τη συνάρτηση. Η καινοτομία σε σχέση με τις δημόσιες προμήθειες και αγορές είναι, έχει ρόλο ιδιαίτερα σημαντικό. Αναφερθήκατε στην ελαστικότητα και απλούστευση που είναι επίσης προτεραιότητες σχετικά με εμά. Είναι μια καλή αφετηρία συνολικά. Πρέπει δυστυχώς να αναφέρω ότι πρέπει να αποχωρήσω. Δεν είναι επειδή είμαι αλλά έχω ανηλυμένες υποχρεώσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ ευχαριστώ. Ο κύριος Κοφέρατη έχει τον λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Επανέρχομαι ε, στην γνωμοδότηση του Στίβεν της πολιτικής μου ομάδας. Ο Στίβεν ε, ταξιδεύει και δεν μπόρεσε να είναι παρόν εδώ και ελπίζω να μην προδώσω, να μην παρεκκλίνω από τη σκέψη του. Προφανώς μιλούμε εδώ για ένα θέμα πάρα πολύ λεπτό και σημαντικό κυρίως για το μέλλον της Ευρώπης. Οι δημόσιες συμβάσεις, όπως το επιθυμεί η Κομισιόν στην Πράσινη Βίβλο, μπορούν να γίνουν ένα εργαλείο πολύ χρήσιμο για την πραγματοποίηση των στόχων της στρατηγικής 2020. Αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει ε, να πληρούνται ορισμένοι όροι και δεν είναι τυχαίο που το ότι η Κομισιόν στην Πράσινη Βίβλο αναφέρει τους όρους αυτούς. Αυτό που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι τα ακόλουθα σημεία. Πρώτο σημείο αναφέρεται στο περιεχόμενο των δημοσίων συμβάσεων. Οι δημόσιες συμβάσεις θα πρέπει να ευνοούν τις ε, ευπρεπείς συνθήκες εργασίας. Υπάρχουν οι κανόνες, οι κανόνες εργασίας του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας και θα πρέπει να αναφέρονται. Ε, το μόνο σημείο το οποίο θα μπορούσε να γίνει ακόμη πιο δεσμευτικό είναι εάν επικαιρώσουμε ε, την σύμβαση του 94 ε, ε, του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Το περιεχόμενο των δημοσίων συμβάσεων θα πρέπει να ενθαρρύνει μια ομοιομορφία στην εργασία, τον σεβασμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων και την ισότητα των όρων προς την ποιότητα της εργασίας. Είναι επίσης σημαντικό ορισμένοι κανόνες, οι οποίοι μέχρι τώρα εφαρμοζόντουσαν με διαφορετικό τρόπο να αναθεωρηθούν και σκέφτομαι τον κανόνα σχετικά με την ανάθεση μιας, ενός έργου με βάση την χαμηλότερη τιμή. Η χαμηλότερη τιμή, η χαμηλότερη προσφορή συνοδεύεται από συστηματική παραβίαση ε, των δικαιωμάτων των ατόμων. Την χαμηλότερη τιμή την επιτυγχάνουμε με κακή ανταμοιβή των εργαζομένων, με κακή εφαρμογή ε, του νόμου και μη τήρηση των ε, κοινωνικών υποχρεώσεων. Θα πρέπει να εξαλείψουμε την ανάθεση ενός έργου με βάση την κατώτερη τιμή και ανταυτού να υπάρχει ένα κριτήριο το οποίο να προσδιορίζεται από την προσφορά, από την, από την πλέον ευνοϊκή οικονομική προσφορά ε, για την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά. Θα πρέπει ε, να ε, μέσα στην διαχείριση των προσφορών, την αντιμετώπιση των προσφορών, θα πρέπει ε, να δούμε ε, ότι πώς θα τηρηθεί ο λόγος, η σχέση δημοσίου-δημοσίου και όχι δημοσίου-ιδιωτικού τομέα. Η σχέση αυτή δημοσίου-δημοσίου επιτρέπει μια σχέση καλύτερη, μια σχέση πιο αποτελεσματική. Και επιτρέπει να καλυφθούν οι προτεραιότητες που ανέφερα και που μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Βεβαίως υπάρχουν και κάποιες δεσμεύσεις ε, οι οποίες ε, συνδέονται και με τις πραγματικές συνθήκες αλλά και με τα δικαιώματα των εργαζομένων. Επίσης δεσμεύσεις οι οποίες συνδέονται με τον σεβασμό ε, των περιβαλλοντικών παραμέτρων. Επομένως η βιωσιμότητα, η αηφορία θα πρέπει να γίνει μία συνιστόσα η οποία θα πρέπει να είναι πάντα παρούσα σε αυτές τις δημόσιες, στους δημόσιους ε, διαγωνισμούς και τις δημόσιες συμβάσεις. Επίσης, ε, η δημόσια σύμβαση θα πρέπει να είναι συνδεδεμένη και με το ίδιο το αντικείμενο της ε, δραστηριότητας και αν μπορεί να δημιουργήσει νέες δραστηριότητες και σε γειτονικέ περιοχές ακόμα καλύτερα. Αλλά ε, θα πρέπει να μην γίνει επικίνδυνη η ίδια η δημόσια σύμβαση εάν ε, οι πρώτερες συνθήκες γίνονται σεβαστές. Επίσης, μιλάμε για δημόσιες συμβάσεις, μιλάμε για δημόσιους διαγωνισμούς. Όμως δεν πρέπει να ξεχνούμε δύο στοιχεία. Το ένα αφορά την ε, αξιολόγηση του χρόνου δηλαδή, ας πούμε, του χρόνου που εγώ έχω ε, χρησιμοποιήσει για να μιλήσω. Γιατί ξέρετε, αλλάζουν οι αρχικές τιμές. Και δεύτερον, η δημιουργία ε, των αλυσίδων αυτών που από την σύμβαση, ε, την κεντρική σύμβαση και την κεντρική εργολαβία προχωράει στην υπεργολαβία. Ε, και ξέρουμε ότι αυτή η επέκταση αυτής της αλυσίδα είναι σχεδόν αυτόματη. Θα πρέπει να το δούμε λίγο αυτό. Σε ευχαριστώ, συνάδελφε. Κύριε ο κύριος Κρόισμαν. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να καλύψω αυτά που ίσως μακρηγόρησε προηγούμενα ο συνάδελφος. Θα είμαι σύντομος. Θέλω να ευχαριστήσω διότι έχουμε ένα πολύ καλό σχέδιο γνωμοδότησης για τον εξυγχρονισμό των δημόσιων συμβάσεων. Οι πιο σημαντικές αρχές των δημόσιων συμβάσεων είναι η διαφάνεια, ο ανταγωνισμός και η μη διακριτική μεταχείριση. Όποιος ακολουθεί αυτές τις αρχές μπορεί να είναι υπεύθυνο και αποτελεσματικός σε σχέση με τη χρήση των κονδυλίων των φορολογουμένων όταν έχουμε δημόσιες συμβάσεις. Αυτό αφορά και τους ε, στόχους που πρέπει να, ακολουθεί, να ακολουθούν. Αυτή η πτυχή ίσως περισσότερο μπορεί να τονιστεί. Συμφωνώ ότι οι διαδικασίες ε, δημόσιων συμβάσεων πρέπει να απλουστευθούν και να καθοριστούν πιο επακριβώς και να διευκολυνθεί η δυνατότητα πρόσβασης σε σχέση με τα, τα διάφορα κοινωνικά στρώματα. Είναι σημαντικές και οι παρατηρήσεις του προλαλήσαντος σε σχέση με την αντική μεταχείριση. Στόχος της στρατηγικής του 2020 είναι ήδη μέσα στα σημερινά πλαίσια να μπορούν οι αρχές να κάνουν περισσότερη χρήση αυτών των δυνατοτήτων, ενώ σήμερα δεν τις χρησιμοποιούν τόσο πολύ. Σαφείς κανόνες θα, θα βελτίωναν την κατάσταση θα οδηγούσαν σε βελτιώσεις. Επίσης η αποτελεσματικότητα και η εξοικονόμηση όσον αφορά τις αγορές πρέπει να συνδέεται με το αντικείμενο αυτό και τις προαναφερθήσεις αρχές που πρέπει να τηρούνται. Μία προώθηση της, προ... της καινοτομίας είναι σκόπιμη και πρέπει να μην παρεκκλίνουν από τις ε, γενικότερες αρχές αυτή τη στιγμή πρέπει να μπορέσουν να εγκριθούν ε, τέτοιου είδους δράσεις. Θα είχαμε περισσότερο καινοτόμε δυνατότητες που θα προσφέραμε. Σε σχέση με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να προσέξουμε η παρακολούθηση πολιτικών στόχων σε σχέση με την εκτέλεση του έργου δεν πρέπει να επιβαρύνει γραφειοκρατικά επιπρόσθετα. Για παράδειγμα, ακριβές πιστοποιήσεις ή πιστοποιητικά θέλουμε πάντα να βοηθάμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και λέμε ότι πάντα τις βοηθάμε. Όταν έρχεται η ώρα χειροπιαστά να το αποδείξουμε, το αμελούμε όμως αυτό. Στις δημόσιες συμβάσεις πρέπει πάντα να θυμόμαστε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επίσης για το e-procurement, τις ηλεκτρονικές μέσω διαδικτύου ε, παραγγελίες. Οι Πορτογάλοι είναι επικεφαλής πρωτοπόροι, 75% γίνεται ηλεκτρονικά στην Πορτογαλία και μεγάλο ποσοστό διοικητικού κόστους εξοικονομείται. Είναι μια πολύ καλή ενδιαφέρουσα λύση που μακροπρόθεσμα θα βοηθήσει και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ευχαριστώ. E Σε ευχαριστώ πολύ και τελευταίος ο συνάδελφός μας ε, Φάβερ. Παρακαλώ σύντομα και εσείς, ε, γιατί έχουμε ψηφοφορίες που ακολουθούν. Σας ευχαριστώ, και τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Σε σχέση με τις δημόσιες συμβάσεις ε, θέλω να πω το εξής. Ε, υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό στα πλαίσια αυτών των ε, δημοσίων συμβάσεων. Τουλάχιστον στην τσεχική δημοκρατία εμείς αντιμετωπίζουμε τη δυσκολία αυτή. Δηλαδή περίπου 10% αυτών των δημοσίων συμβάσεων, το 10% εξαφανίζεται, εξανεμίζεται σε διαφθορά, λαδώματα κτλ. Ε, Επομένω, νομίζω ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα και για την προστασία ε, των συμβάσεων κατά αυτή την έννοια. Σε ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν η συνάδελφό μα, ε, Julie Γκέρλινγκ θέλει ακόμα να πει κάτι. Θέλετε να παρέμβετε για να ολοκληρώσετε τη συζήτηση αυτή. Yes, thank you. Thank you, Chairman. I know you want to get on. Ναι, Πρόεδρε, ξέρω ότι θέλετε να προχωρήσετε στην ψηφοφορία. Ε, γι' αυτό λοιπόν δεν θέλω να μακρηγορήσω. Ε, νομίζω ότι ούτως ή άλλως ε, θα είναι μια σύντομη γνωμοδότηση, μικρή γνωμοδότηση και θα έχουμε και την ανταλλαγή απόψεων με τους σκιώδεις συγητές. Παρ' όλα αυτά να κάνω κάποια σχόλια. Πολλοί ομιλητές ε, έθιξαν το θέμα των περιβαλλοντικών κριτηρίων. Είμαι μέλος και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και εκεί συντάσσουν γνωμοδότηση ε, επομένως νομίζω ότι θα πρέπει να αφήσουμε αυτά τα στοιχεία που αφορούν το περιβάλλον. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να περιορίσουμε τα σχόλιά μας σε αυτά που είναι αρμοδιότητα ε, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, τα, ε, της Επιτροπής Απασχόλησης. Τα σχετικά με την Επιτροπή Περιβάλλοντος θα τα περιλάβει η γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα τα ελέγξω θα ελέγξω όλα τα στοιχεία και θα δούμε ε, ε, ε, επίσης το θέμα των παραχωρήσεων και αυτό θα το ελέγξω. Υπάρχουν, αναφέρθηκαν και κάποια άλλα σχόλια με τα οποία δεν μπορώ να πω ότι διαφωνώ ε, τρομερά. Πάντω, αυτό που μπορώ να πω είναι να είμαστε, ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί έτσι ώστε να μην παρισφρήσουν πολιτικά ε, στοιχεία. Κυρίως ε, εάν μιλάμε για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την ανάμειξή του και την δυνατότητα συμμετοχής τους στις δημόσιε συμβάσεις. Θα υπάρξουν βέβαια φαντάζομαι και τροπολογίες. Και όπως ε, ε, σας είπα, σας ξαναλέω ότι ε, θα συζητήσω και με τους σκιώδεις και οτιδήποτε χρειάζεται θα το διευθετήσω. Με ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Η περίοδος για την κατάθεση τροπολογιών, η κατάθεση θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 23 Ιουνίου το μεσημέρι, 12.00. Μετά θα ψηφιστεί στις 13 Ιουλίου στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή το θέμα και θα αποσταλεί στην, Ολομε... στην, Ευρωπαϊκή Επιτρο... στην Επιτροπή ΙΝΚΟ, με συγχωρείτε, για να εγκριθεί καταρχήν στις 19 Σεπτεμβρίου και θα πάει στην περίοδο Συνόδου Ολομέλειας τον Οκτώβριο στην Ολομέλεια. Ολοκληρώνουμε αυτή μας τη συζήτηση και περνάμε τώρα, αν συμφωνείτε, στην περίοδο ψηφοφοριών, στις ψηφοφορίες. Ελπίζω όλοι να έχετε τις κάρτες σας για να μπορείτε ηλεκτρονικά να ψηφίσετε. Αν δεν τις έχετε, παρακαλώ να υπάρξει μια ειδοποίηση, να, μας το, να το ξέρουμε. Θα ξεκινήσουμε με την έκθεση Άνταμ Κόσα για την κινητικότητα και την ένταξη κοινωνικά των ατόμων με αναπηρίες και την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία 2010-2020. Όλα είναι έτοιμα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι και μπορούμε να ξεκινήσουμε λοιπόν τις ψηφοφορίες μας. Πρώτη παράγραφος, πρώτο εδάφιο. Τροπολογία 56. Με προφορική τροποποίηση του εισηγητή. Όσοι είναι υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. και επίσης προφορική τροποποίηση του εισηγητή μας νομίζω συμπεριλαμβάνεται, όχι. Είναι ξεχωριστή, λέει ο μιλήτης. Υπάρχει μια άλλη λοιπόν προφορική τροποποίηση σε αυτό το εδάφιο του εισηγητή. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. νομίζω θα πρέπει να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά για αυτή την προφορική τροποποίηση. Πέρας ψηφοφορίας. Τριάντα υπέρ, 13 εναντίον, μία αποχή, εγκρίθηκε. Και τώρα η τροπολογία 55 παράγραφος 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Η τροπολογία 11 της Επιτροπής Περιβάλλοντος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 97 έχει αποσυρθεί. Περνάμε στην παράγραφο 2. Συμβιβασμός α. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Καταπίπτουν οι τροπολογίες που ακολουθούν μέχρι την παράγραφο 3. Συμβιβασμός β. Β. Υπέρ. Κατά αποχές. Παρακαλώ να είναι πιο σύντομος ο διερμηνέας γιατί χάνουμε την ακολουθία με τον ρυθμό αυτό. Ah, Σας ευχαριστώ εντάξει. Τρίτη παράγραφος, συμβιβασμός Β, επαναλαμβάνω, ψήφι υπέρ ψήφι κατά αποχές εγκρίνεται καταπίπτουν οι τροπολογίες που ακολουθούν και περνάμε φτάνουμε στην παράγραφο 3α τροπολογία 3 της Επιτροπής Γυναικών ψήφι υπέρ κατά αποχές Przepraszam bardzo, ale my nie mamy polskiego tłumaczenia w ogóle. Nic nie słyszymy w słuchawkach. φαίνεται ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Λοιπόν, με την πολωνική διερμηνία υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Τι είναι. Υπάρχει διερμηνία στα πολωνικά, παρακαλώ. Μπορείτε να μας ειδοποιήσετε αν έχετε διερμηνία στα πολωνικά. Ναι, ναι, ναι, ναι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ακούμε, ακούμε τη διερμηνή. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν. Εντάξει, υπάρχει λοιπόν διερμηνία και θα ξαναξεκινήσουμε. Θα ξαναξεκινήσουμε. Yes. Λοιπόν, ξαναξεκινάμε. Παράγραφος 3α νέα. Τροπολογία υπαριθμών 3 της Επιτροπής Γυναικών. <clears throat> Ψήφι υπέρ. Ε, Ψήφι κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Παράγραφος 4. Συμβιβασμός σε γάμα. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Καταπίπτουν οι υπόλοιπε τροπολογίες μέχρι που φτάνουμε στην παράγραφο 5. Συμβιβασμός ΔΕΛΤΑ. D. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Καταπίπτουν πάλι οι ακόλουθες τροπολογίες μέχρι την παράγραφο 6. Συμβιβασμός ε, ή, υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Και περνάμε στην παράγραφο 6α ε, νέα, τροπολογία 84. Κοφεράτη, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Περνάμε στην τροπολογία 85 του εισηγητή. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Παράγραφος 7. Ε, Συμβιβασμός F. Σίγμα ταφ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Και περνάμε στην παράγραφο 7α νέα Συμβιβασμός G, Z, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Και πάμε στην παράγραφο 7α νέα. Τροπολογία 90. Ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Περνάμε στην παράγραφο 8. Συμβιβασμός ήταν H, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Και πάμε Περνάμε λοιπόν στην παράγραφο 8, στην τροπολογία 95 έχουμε μια τροπολογία της κυρίας Σρότερ εδώ. Η γραμματεία μου λέει ότι θεωρεί ότι το δεύτερο τμήμα μπορεί να ψηφιστεί ως προσθήκη στον συμβιβασμό H. Έτσι θα ψηφίσουμε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Και περνάμε τώρα στο, στην παράγραφο 8α νέα, συμβιβασμός ε, I, e, υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. Και περνάμε στην παράγραφο 8α νέα, τροπολογία 103 του εισηγητή υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Η τροπολογία, στη 182 τροπολογία υπέρ, κατά, απόχες, απορρίφθηκε. Τροπολογία. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά, εντάξει, θα ελέγξουμε. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την 182 τροπολογία της κυρίας Σόρεντερ. Άρχεται η ψηφοφορία. Ε, στα... Πέρας ψηφοφορίας και αποτέλεσμα εγκρίθηκε. Είχατε δίκιο. Εδώ από εδώ δεν το είδαμε. Λοιπόν, εντάξει, εγκρίθηκε η 182. Και έτσι πάμε στην παράγραφο 8α νέα, πάλι τροπολογία 105, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Περνάμε στην παράγραφο 9, συμβιβασμός J, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Και πάμε στην Παράγραφο 9α νέα, τροπολογία 111. Υπέρ, κατά, αποχές. Νομίζω απορρίφθηκε, αλλά πιθανότατα μπορούμε να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Είναι καλύτερο να ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την 111, άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ε, στα... Πέρας ψηφοφορίας τώρα. Πράγματι απορρίφθηκε η τροπολογία αυτή. Μετά έχουμε την παράγραφο 10. Συμβιβασμός K. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Συμβιβασμός L. Στην παράγραφο 11. Υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε και περνάμε στην παραγραφό 11 ναι, ε, την τροπολογία 118 έχουμε. Μπορούμε να την ψηφίσουμε ως προσθήκη την 118. Ψήφι υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι απορρίφθηκε, αλλά θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την 118 τροπολογία. Ε, Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα εγκρίθηκε. Και στην παράγραφο που έχουμε 11α, τροπολογία 121 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε η 121. Περνάμε στην παράγραφο 12. Συμβιβασμός M υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Πάμε τώρα στον συμβιβασμό, όχι, στην τροπολογία 129, στην παράγραφο 13, 129 του εισηγητή, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Και πάμε στο, στην παράγραφο 14. Συμβιβασμός εν υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Και έτσι περνάμε στην παράγραφο 14. Έχουμε την τροπολογία 136 και την 137 στην 14α. Είναι ταυτόσιμες. Ψήφοι υπέρ αυτών κατά αποχές εγκρίθηκαν. Και πάμε στην παράγραφο 15. Τροπολογία 139. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 140. Ψήφι υπέρ. Κατά. Θα επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά αν θέλετε. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την 140. E Ψηφίζουμε την 140. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα. Ισοψηφία. 23 υπέρ 23 εναντίον. Απορρίφθηκε λοιπόν σύμφωνα με τον κανονισμό λόγω ισοψηφίας. Τροπολογία 141 του εισηγητή. Υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίθηκε. Η... Μπορούμε να ψηφίσουμε την 142 που είναι συμβατή και αυτή. Ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Περνάμε στην παράγραφο 15α νέα, τροπολογία 143, υπέρ, κατά, απόχες, εγκρίθηκε. 144, υπέρ, κατά, απόχες, εγκρίθηκε. 145, υπέρ, κατά, απόχες. Νομίζω ότι απορρίφθηκε. Παρακαλώ, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε την 145. Πέρα Πέρας ψηφοφορίας. Πέρας ψηφοφορίας, μάλιστα. Εγκρίθηκε με μία ψήφο διαφορά. 24 υπέρ, 23 εναντίον. Εγκρίθηκε. Περνάμε στην 146 τώρα. Με προφορική τροποποίηση του εισηγητή. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Περνάμε στην... Ναι, παρακαλώ, έχετε τον λόγο κυρία Σρέντερ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Υπάρχει προφορική τροποποίηση για την τροπολογία 147. Δεν θέλουμε να εγκριθεί η προφορική τροποποίηση. Θέλουμε το αρχικό κείμενο να ψηφιστεί χωρίς προφορική τροποποίηση. Πρόεδρος, Βλέπω ότι υπάρχει αντίρρηση λοιπόν στην προφορική τροποποίηση, δεν θα ψηφιστεί. Παραμένει το αρχικό κείμενο στο οποίο θα ψηφίσουμε λοιπόν. Πολύ καλά. Και περνάμε ακριβώς στην, τροπολογία 15 της Επιτροπής Γυναικών. Ε, συγγνώμη. Ναι, ζητώ συγγνώμη η 147 στο αρχικό κείμενο, χωρίς την προφορική τροποποίηση, όπως πρότεινε ακριβώς η κυρία Σρότερ υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίθηκε η 147. Και τώρα μάλιστα μπορούμε να περάσουμε στην Επιτροπή Γυναικών. Τροπολογία 11. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Και περνάμε στην παράγραφο 16. Συμβιβασμός ο, ομικρον, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε η συμβιβαστική τροπολογία. Και περνάμε στην παράγραφο 16α νέα, τροπολογία 156. Ψήφι περ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Τροπολογία 158. Και εδώ πάλι με προφορική τροποποίηση. Και έχουμε ακόμα και μια πρόταση του εισηγητή μετά την παράγραφο 31 δηλαδή ψήφι υπέρ κατά άποχες εγκρίθηκε περνάμε στην παράγραφο 17 τροπολογία 159 του εισηγητή υπέρ κατά άποχες εγκρίθηκε τροπολογία 160 ψήφι υπέρ κατά άποχες εγκρίθηκε 161 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 162 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε είναι η καθυστέρηση λόγω διερμηνίας λέγεται στην Πρόεδρο 163 και η τροπολογία 167 είναι ταυτόσιμες ψηφίζουμε από κοινού υπέρ αυτών κατά αποχές εγκρίθηκαν και περνάμε στην τροπολογία 164 και με προφορική τροποποίηση του εισηγητή που ε, αναφέρεται στο κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 100 τροπολογίες 168 και συνεχείς ακόλουθες καταπίπτουν. Περνάμε στην 169. 165 διορθώνει η πρόεδρος. Ζητώ συγγνώμη 165 λέει η πρόεδρος. 165 τροπολογία. Μάρα Μπισότο. Στην παράγραφο 18, εδάφια 18. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Θα ήθελα να υπαλληθεύσουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε την 165 τροπολογία. Άρχεται η ψηφοφορία λοιπόν. Τώρα πέρας ψηφοφορίας. Α, ένα μέλος του ΕΛΚ παραπάνω συμμετέχει στην ψηφοφορία. Ένα μέλος του ΕΛΚ ψηφίζει και είναι παραπάνω. Εντάξει, αποσύρθηκε η ψήφος παραπάνω. Πέρας ψηφοφορίας τώρα. Εγκρίθηκε η τροπολογία αυτή. Είναι σαφές. 28 ψήφοι υπέρ, 17 εναντίον. Επαρκεί και εγκρίθηκε. Λοιπόν, περνάμε στην τροπολογία 169. Πιστεύω ότι 166 κατέπεσε. Σωστό. Εντάξει. Περνάμε στην 169. Επειδή 166 κατέπεσε λοιπόν. 169 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 170 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 172 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε αν υπάρχουν αμφιβολίες να επαναλάβουμε λοιπόν άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά γιατί υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες ψηφίζουμε την 172 άρχεται η ψηφοφορία λοιπόν Πέρας ψηφοφορίας τώρα. Αποτέλεσμα εγκρίθηκε 32 υπέρ, 13 εναντίον. Εγκρίθηκε. Περνάμε στην 173. Υπέρ. Κατά. Απόχες. Απορρίφθηκε. Από το Προεδρείο δεν υπάρχουν αμφιβολίες. Απορρίφθηκε. 174 του εισηγητή ψήφι κατά, αποχές, απορρίφθηκε. Θέλετε να επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά, μάλιστα, άρχεται η ψηφοφορία, ψηφίζουμε την 174 στην παράγραφο 19, τροπολογία του εισηγητή. πέρας ψηφοφορίας Πράγματι απορρίφθηκε. 25 εναντίον και 20 υπέρ. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 175. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 176, καταπίπτει 176 και περνάμε στην 177, παράγραφος 19α νέα. 177 Λίσια Ροζόλη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 178. Υπέρ. Κατά. Θα επαναλάβουμε την ψηφοφορία. Ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε την 178. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας τώρα. «29 υπέρ, 17 εναντίον». Εγκρίθηκε λοιπόν. Και περνάμε στην 170... 180 ε, επίσης, 181 κατέπεσε και αυτή. Περνάμε στην παράγραφο 21 τροπολογία 184 υπέρ κατά άποχες εγκρίθηκε τροπολογία 185 ναι παρακαλώ εσείς έχετε τον λόγο ψηφίσαμε την 180 ερώτηση Α, ah, sí. Μάλιστα έχετε δίκιο, έχετε δίκιο, διότι 180 είναι συμβατή πράγματι με την προηγούμενη. Σωστό και σας ευχαριστώ για την παρατήρηση συνάδελφε. Θα ψηφίσουμε την 180 τροπολογία τώρα λοιπόν. Κίνγκε Γκόντσε, ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Και τώρα μάλιστα μπορούμε να περάσουμε στην 184. Ψήφι υπέρ της 184. Και την 181 λέτε. Να την ψηφίσουμε και αυτήν. Εντάξει. Λοιπόν, λοιπόν περνάμε. Ναι, μου είπε η γραμματεία ότι έχουν καλυφθεί οι προηγούμενες. Η 186 απομένει, περνάμε στην 186. Ψηφίζουμε την 186 υπέρ κατά αποχές νομίζω απορρίφθηκε αλλά καλύτερα να υπαλληθεύσουμε ηλεκτρονικά υπάρχουν αμφιβολίες ψηφίζουμε την 186 άρχεται η ψηφοφορία 186 τροπολογία πέρας ψηφοφορίας τώρα εγκρίθηκε και περνάμε στον συμβιβασμό π. Στην παράγραφο 22. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Και έτσι θα περάσουμε τώρα. Οι άλλες τροπολογίες καταπίπτουν. Περνάμε στην 194 τροπολογία. Παράγραφος 22α νέα. Ψήφι υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίθηκε. 196 με προφορική τροποποίηση Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Περνάμε στην παράγραφο 23. Έχουμε τον συμβιβασμό Q. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο, κύριε Σιγητά. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να επιστήρωσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι μετά από την χτεσινή μας ε, συζήτηση με τους συναδέλφους του ΕΛΚ ε, φτάσαμε σε ένα συμβιβασμό και συστήνω οι συνάδελφοί μου στο ΕΛΚ να στηρίξουν το συμβιβασμό αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ καλά. Θα ψηφίσουμε λοιπόν την παράγραφο 23, τον συμβιβασμό Q. Υπέρ λοιπόν, κατά αποχές εγκρίθηκε. καταπίπτουν οι ακόλουθες οι υπόλοιπες τροπολογίες. Φτάνουμε μέχρι την τροπολογία, πιστεύω, 204, έτσι. 204 τροπολογία. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Περνάμε στην τροπολογία, στην παράγραφο 23β. Έχουμε το συμβιβασμό R. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Καταπίπτουν οι υπόλοιπε τροπολογίε. Φτάνουμε μέχρι το συμβιβασμό S στην παράγραφο 24. Υπέρ. Συμβιβασμό S. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Και περνάμε τώρα. Καταπίπτουν οι υπόλοιπε τροπολογίε μέχρι την τροπολογία 214. Στην παράγραφο 24α νέα. Τροπολογία 214 υπέρ Κατά. 214 τροπολογία, παρακαλώ. Στην σελίδα 25 του δικού μου κατάλογου ψηφοφορίας. 214 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Περνάμε στην παράγραφο. Στην τροπολογία 216 λοιπόν. Υπέρ κατά άποχες απορρίφθηκε νομίζω η 216 πάμε στην 217 υπέρ κατά άποχες απορρίφθηκε όχι λέτε όχι Ωραία. Μπορούμε να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την 217. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ε, βατου... Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. 23 εναντίον, 21 υπέρ. Λοιπόν, περνάμε στην 219 τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Απόχες. Απορρίφθηκε. Πάμε στην 223 με προφορική τροποποίηση, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Παράγραφος 25 τώρα, τροπολογία 224, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 225, είναι συμβατή αυτή, ψήφι υπέρ, κατά, απόχες εγκρίθηκε 226 υπέρ κατά απόχες εγκρίθηκε 229 υπέρ κατά πρέπει να ελέγξουμε ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά ψηφίζουμε την 229 τροπολογία άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίθηκε 23 ψήφοι υπέρ 21 εναντίον. Και περνάμε στην 231 τροπολογία. Υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίθηκε. 232 υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίθηκε. 233 υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίθηκε. Η 236 αποσύρθηκε. Περνάμε στην παράγραφο 26, παρά, ε, συμβιβασμός ε, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Και περνάμε στην παράγραφο έχουμε την τροπολογία 239 ωστόσο στην παράγραφο 26 239 παράγραφος 26 ως προσθήκη αυτή η τροπολογία έτσι, στο συμβιβασμό προσθήκη υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Μπορούμε να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την 239 ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας απορρίφθηκε 27 εναντίον 19 υπέρ. Περνάμε στην παράγραφο 27. Συμβιβασμός U. Ψήφι υπέρ του συμβιβασμού U. Υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Πάμε στην παράγραφο 27, τροπολογία 245, με προφορική τροποποίηση 245, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Παράγραφος 28, συμβιβασμός Β, υπέρ κατά απόχες εγκρίθηκε και περνάμε οι υπόλοιπες καταπίπτουν φτάνουμε στην τροπολογία 250 στην παράγραφο 28α νέα στη σελίδα 28 250 τροπολογία ψήφι υπέρ κατά απόχες εγκρίθηκε 251 251 λοιπόν υπέρ κατά αποχές νομίζω απορρίφθηκε αλλά θα ελέγξουμε υπάρχουν αμφιβολίες νομίζω όχι έτσι ε λοιπόν περνάμε στην 255 ψήφι υπέρ 255 τώρα με προφορική τροποποίηση ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε Ανθρωπολογία 256. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε και περνάμε στην παράγραφο 29. Συμβιβασμός W. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Και περνάμε στην παράγραφο 29 τροπολογίες 261-291 είναι ταυτόσιμες, μπορούν να ψηφιστούν από κοινού υπέρ αυτών κατά αποχές εγκρίνονται. Περνάμε στην 262 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 263 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε και περνάμε στην 264. Έχουμε εδώ και προφορική τροποποίηση του εισηγητή υπέρ, κατά, απόχες, εγκρίθηκε. Περνάμε στην 265, υπέρ, κατά, απόχες, εγκρίθηκε. 200... Όχι λέτε, δεν είχαμε διαρμηνία για αυτή την ψήφιση και έτσι πρέπει... Λοιπόν, θα επαναλάβουμε την ψηφοφορία γιατί, για το θέμα αυτό της διαρμηνίας σε κάποιες γλώσσες. Τροπολογία 265 στην παράγραφο 30. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Και περνάμε τώρα λοιπόν στην τροπολογία 266 και επίσης 267 που και οι δύο μπορούν να ψηφιστούν από κοινού είναι ταυτόσιμες ψήφοι υπέρ αυτών κατά αποχές εγκρίθηκαν και περνάμε στην τροπολογία 268 με τροπολογία του εισηγητή τροποποίηση υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε Περνάμε στην τροπολογία. 269. Ήρντα Φιγκερέντο λοιπόν, υπέρ. Κατά. Απόχες. Νομίζω εγκρίθηκε, αλλά θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία, ψηφίζουμε την 269. Ε, Πέρας ψηφοφορίας. 23-23 ισοψηφία. Απορρίφθηκε λοιπόν. Μάλιστα. Τροπολογία 270. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 272. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 271. Υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 273 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε δεν υπάρχουν αμφιβολίες ε. λοιπόν 200, 275 με προφορική με τροποποίηση του εισηγητή ψήφι υπέρ κατά απόχες εγκρίθηκε 276 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε περνάμε τώρα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος τροπολογία 14 Επιτροπής Περιβάλλοντος ένβη υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε Πάμε στην, στην παράγραφο 31, τροπολογία 277 του εισηγητή. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Τροπολογία 279, με προφορική τροποποίηση του εισηγητή. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Περνάμε στην τροπολογία NV3. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. NV20, υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. Πάμε στην τροπολογία 280 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 281 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 282 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 283 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 284 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 285 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 286 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 287 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 288 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 289 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 290 και 291 είναι ταυτόσιμες ψηφίζουμε όχι όχι δεν είναι λοιπόν ταυτόσιμες ζητώ συγγνώμη μάλιστα το είδα λοιπόν παράγραφος 36 θα ψηφίσουμε την τροπολογία 290 εδώ υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε η 291 είναι συμβατή με την προηγούμενη αλλά ξεχωριστά θα την ψηφίσουμε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Όμως έχω κάποιες αμφιβολίες και θα ήθελα να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την 291, άρχεται η ψηφοφορία. Ε, ε... Πέρας ψηφοφορίας. Πέρας ψηφοφορίας λοιπόν. Αποτέλεσμα 22 εναντίον, 21 υπέρ. Καταψηφίστηκε, απορρίφθηκε. Τροπολογία 293. Μπορούμε να ψηφίσουμε από κοινού 293, 94, 95, 96, 97, 98, όλες αυτές από κοινού. Μπορούμε να ψηφίσουμε ομού, ψήφι υπέρ αυτών. Κατά, αποχές, εγκρίθηκαν. Και περνάμε στην τροπολογία, στο, στην παράγραφο 36, το προφορική τροποποίηση έχουμε στην τροπολογία αυτή, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Και περνάμε επίσης τώρα στις αιτιολογικές σκέψεις. Στο α, τροπολογία 17, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. Η τροπολογία 18, υπέρ, κατά αποχές απορρίφθηκε. Όχι, εγκρίθηκε, ζητώ συγγνώμη λέει η πρόεδρος. Η δεύτερη αυτή τροπολογία Β εγκρίθηκε. Περνάμε στην αιτιολογική σκέψη Β. Ε, συμβιβασμός εξ υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Και περνάμε στην τροπολογία 24. Ψήφι υπέρ κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Νομίζω εγώ, αλλά θα ελέγξουμε αν θέλετε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία, ψηφίζουμε την 24. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε, όπως είχα προαναφέρει, 24 υπέρ, 21 εναντίον. Η τροπολογία 33 τώρα. Κατέπεσε αυτή. Ωραία. Και περνάμε NVE τροπολογία, NVE, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. 25 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε και περνάμε στον συμβιβασμό C. Όχι, συγγνώμη, στην αιτιολογική σκέψη C, συμβιβασμός Y. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. Αιτιολογική σκέψη D, συμβιβασμός Z. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Καταπίπτουν οι υπόλοιπε τροπολογίες γι' αυτό, για το, την αιτιολογική σκέψη D. Ε, πάμε στην τροπολογία 32, αιτιολογική σκέψη D, α, νέα. 32, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Τροπολογία 34 τώρα, υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 46. Καταπίπτει αυτή. Επίσης καταπίπτει και η 50. Τροπολογία 50. Μάλιστα. Και έτσι περνάμε στην αιτιολογική σκέψη Ι. E. Συμβασμός ΑΑ. AA. Υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίθηκε. Περνάμε τώρα στην NVF. Τροπολογία NVF. Επιτροπής Περιβάλλοντος. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε, νομίζω. Δεν υπάρχουν αμφιβολίες. Υπάρχουν. Εφόσον υπάρχουν πρέπει να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Λοιπόν, NVF. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας τώρα. Αποτέλεσμα 20 υπέρ 24 εναντίον καταψηφίστηκε. Απορρίφθηκε λοιπόν. Και περνάμε τώρα στον συμβιβασμό BB. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Και πάμε τώρα στην αιτιολογική σκέψη F. Τροπολογία 41. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 42. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. Προφορική τροποποίηση του εισηγητή τώρα. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Πάμε στην τροπολογία 43 υπέρ κατά άποχες εγκρίθηκε. Πάμε τώρα στην 44 που είναι συμβατή υπέρ κατά άποχες εγκρίθηκε. Επίσης η 45 είναι και αυτή συμβατή υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα, θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την 45, άρχεται η ψηφοφορία, στην αιτιολογική σκέψη H. Πέρα τώρα. 27 υπέρ, 17 εναντίον. Έτσι εγκρίθηκε λοιπόν. Και περνάμε τώρα στην NVI ε, συγγνώμη, η προφορική τροποποίηση είναι NVI, με προφορική τροποποίηση υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 47, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. 48, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. 49, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. 51, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. 53, υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε 52 όχι η 52 καταπίπτει καταπίπτει μια και εγκρίθηκε η 53 εντάξει και περνάμε στην τροπολογία Επιτροπής Αναφορών 1 ΠΕΤ 1 με προφορική τροποποίηση υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε Επιτροπής Αναφορών η 2 με προφορική τροποποίηση υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε και περνάμε τώρα στα σκεπτικά Envy, SIT, τροπολογία 3. Έχουμε το πρώτο σκεπτικό υπέρ κατά αποχές. Εγκρίθηκε με την προφορική τροποποίηση. Περνάμε στις τροπολογίες 1 και 2 πρώτα, που είναι ταυτόσιμες. Υπέρ αυτών κατά αποχές. Εγκρίθηκαν. Περνάμε στην Envy Sit 1. Τροπολογία Envy Sit 1. Υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Περνάμε στην συστροπολογής 3 και 4. Είναι ταυτόσιμες υπέρ αυτών. Κατά αποχές εγκρίθηκαν. Η τροπολογία 5 τώρα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Και η τροπολογία 6. 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Θέλετε να ελέγξουμε. Όχι. Εντάξει, εγκρίθηκε. Δεν υπάρχουν αμφιβολίες. Οι τροπολογίες 7 και 8 είναι ταυτόσιμες. Ψηφίζουμε υπέρ αυτών. Κατά αποχές εγκρίθηκαν. Επίση η τροπολογία 9 υπέρ. Τροπολογία 9 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Περνάμε στο σκεπτικό 11. Προφορική τροποποίηση εδώ του εισηγητή. Ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Στο σκεπτικό 13 τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Πάμε στην τροπολογία 13. 13 στο σκεπτικό 16 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Πάμε στις τροπολογίες 11 και 12 που είναι ταυτόσιμες υπέρ αυτών κατά αποχές εγκρίθηκαν. Περνάμε στις τροπολογίες 14 και 15 που και αυτές είναι ταυτόσιμες. Υπέρ αυτών, κατά, αποχές, εγκρίθηκαν. Εγκρίθηκαν, σωστό. Η 16 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Ε, Εδώ η γραμματεία μόλις μου είπε ότι θα έπρεπε να έχουμε μια αποκοινού ψήφιση όλων των τροπολογιών που είναι προφορικές ε, τροποποίησεις από το 17 σκεπτικό 17 17α νέο του εισηγητή μέχρι όλες τις τροπολογίες τις προφορικές με προφορική τροποποίηση μέχρι το τέλος των προφορικών τροποποίησεων του εισηγητή μέχρι την NV SIT 8 όλες λοιπόν υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκαν. Και περνάμε λοιπόν έτσι στο σκεπτικό 17 έχουμε την NVC 7 της Επιτροπής Περιβάλλοντος υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε Ξαναγυρίζουμε στην προφορική τροποποίηση. NVC το 8. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. NVC 11. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. NVC 12. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. NVC 13. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Και πάμε τώρα στην τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά βέβαια. Άρχεται η ψηφοφορία, τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Έχουμε 46 που συμμετείχαν στην ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας λοιπόν. 42 ψήφοι υπέρ, 3 εναντίον και μία αποχή. Συγχαρητήρια στον εισηγητή μας. Και τώρα μπορούμε να περάσουμε λοιπόν στην ψήφιση της έκθεσης Ουγγουρεάνου η προαγωγή της ελευθερίας κυκλοφορίας των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, η πρώτη τροπολογία Είμαστε σε θέση να ξεκινήσουμε και να ψηφίσουμε. Ξεκινάμε λοιπόν. Τροπολογία 26 στην παράγραφο 1 νέα. Παράγραφος 1 νέα υπέρ 26 κατά απόχες. Νομίζω εγκρίθηκε. Αλλά αν υπάρχει αμφιβολία άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά θα ελέγξουμε. Ψηφίσουμε την 26. Shut up the sound. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Ε, Πάμε, Λίμπε 9, τροπολογία Λίμπε 9, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε και αυτή. Στην παράγραφο 2, τροπολογία 27, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. Συμβιβασμός Α υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. πίπτη 28 και περνάμε στην Επιτροπή Γυναικών 17. Τροπολογία 17 Επιτροπής Γυναικών υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 29 τροπολογία υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Τροπολογία 30 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Λιμπ 5 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Η τροπολογία 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Επιτροπής γυναικών 12 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Επιτροπής γυναικών 18 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε η τροπολογία 32 υπέρ κατά αποχές νομίζω απορρίφθηκε λίμπε 6 υπέρ λίμπε 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Επιτροπή Γυναικών 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 33 σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές Απορρίφθηκε το δεύτερο τμήμα. Γυναικών 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 36 υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε Επιτροπής Γυναικών 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 38 υπέρ κατά Έχω κάποιες αμφιβολίες. Προτιμώ να επαληθεύσουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Τροπολογία 38. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Λίμπε 15. Σε δύο τμήματα. Όχι. Με προφορική τροποποίηση μόνο. Εντάξει. Λίμπε... Γίνεται δεκτή. Είναι δεκτή η προφορική τροποποίηση. Ωραία. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε με την προφορική τροποποίηση. Εντάξει. 39 τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Απορρίφθηκε μάλιστα. Επιτροπής γυναικών η 4. Υπέρ. Κατά. Συγγνώμη, αλλά δεν ήταν σαφές το αποτέλεσμα. Λοιπόν, θα επαναλάβουμε. Η Επιτροπή Γυναικών, η Πρωτοπολογία 4, υπέρ Μάλιστα, τώρα είναι σαφέστερο. Κατά αποχές εγκρίθηκε λοιπόν. Ωραία. Τροπολογία 40. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. Λίμπε 10. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Η 41. Υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε η Λίμπε 24 υπέρ κατά εγκρίθηκε αποχές εγκρίθηκε η 42 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε δεύτερο τμήμα υπέρ κατά απορρίφθηκε αποχές απορρίφθηκε το δεύτερο τμήμα Επιτροπής Γυναικών 5 υπέρ, πάλι σε δύο τμήματα, συγγνώμη, Επιτροπής Γυναικών 5, το πρώτο τμήμα πρώτα, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε, δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε το δεύτερο τμήμα. Η 43 καταπίπτει και περνάμε στην παράγραφο 8, συμβιβασμός B, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Πάμε τώρα στην Τροπολογία 48 υπέρ κατά αποχές κατά αποχές εγκρίθηκε 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε η τροπολογία 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε περνάμε στο συμβιβασμό C γάμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε Πάμε στην τροπολογία 53. Οι άλλες καταπίπτουν οι προηγούμενες. Υπέρ της 53. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε η 53. Πάμε στην 54. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Πάμε στην 55. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Η τροπολογία 56 τώρα. Υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε εγκρίθηκε συγγνώμη ζητώ συγγνώμη εγκρίθηκε η 56 Θέλετε να επαναλάβουμε την ψηφοφορία. Εγκρίθηκε η 56, εγκρίθηκε. Εντάξει. Τροπολογία 57 τώρα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Λίμπε 1. Έχουμε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Δεν βλέπω πώς ψηφίζεται. Θα ήθελα να υπαλληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία στο δεύτερο τμήμα της ΛΥΜΠΕ 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Ε, Πέρας ψηφοφορίας. 18 υπέρ, 21 εναντίον, 2 αποχές, απορρίφθηκε. Ε, και περνάμε τώρα. Επιτροπή γυναικών 1, τροπολογία 1, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. Πάμε στην τροπολογία 58 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Τροπολογία 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Η 60 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές Απορρίφθηκε το δεύτερο τμήμα. Πάμε στην τροπολογία 61. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Η τροπολογία 62. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε η 62. Για την 62 πιστεύω ότι εγκρίθηκε. Λοιπόν, να επαναλάβουμε. Ψηφίζουμε την 62. Τροπολογία 62. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Δεν υπήρχαν αμφιβολίες για μένα, αλλά τέλος πάντων ελέγχουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Μάλιστα 39 υπέρ. Σαφέστατο το αποτέλεσμα. Υπερψηφίστηκε. Για μένα ήταν σαφές. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Θα ψηφίσουμε τώρα. Λίμπε. Λίμπε 12. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε νομίζω δεν υπάρχουν αμφιβολίες διαμαρτυρίες εντάξει ωραία θέλετε να ελέγξουμε ελέγχουμε ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα της ΛΥΜΠΕ 12 άρχεται η ψηφοφορία Πέρας ψηφοφορίας. 25 υπέρ, 17 εναντίον. Εγκρίθηκε. Μάλιστα, σωστό. Λίμπε 13. Λίμπε 13 υπέρ. Κατά. Λοιπόν, θα ελέγξουμε για την Λίμπε 13, διότι δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα πώς ψηφίζουν οι ομάδες. Λίμπε 13, άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. ...25 υπέρ, 16 εναντίον, εγκρίθηκε. Και περνάμε στην τροπολογία 63, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 64 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 66 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε απορρίφθηκε μάλιστα. Η 67 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε το δεύτερο τμήμα. Τροπολογία 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Η 69 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Περνάμε στην παράγραφο 12. Συμβιβασμός δι υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Περνάμε στην ΛΥΜΠΕ 25, τροπολογία ΛΥΜΠΕ 25, υπέρ, κατά. Κατά. ΛΥΜΠΕ 25, κατά. Αν υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες, άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. ΛΥΜΠΕ 25. Ε, Άρχεται η ψηφοφορία, ψηφίζουμε την ΛΥΜΠΕ 25 τροπολογία. Ε. Πέρας ψηφοφορίας. Πέρας ψηφοφορίας. 13 υπέρ 25 εναντίον απορρίφθηκε. Η 72 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. Η 73 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε η 74 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε η 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε η 76 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε η 77 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Νομίζω εγώ ότι απορρίφθηκε. Όχι, εντάξει. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά, έρχεται η ψηφοφορία. Εντάξει, θα ψηφίσουμε την 77 ηλεκτρονικά. Άρχεται. Ε, Πέρας ψηφοφορίας. εγκρίθηκε η 78 καταπίπτει η 78 η 79 υπέρ κατά απόχες απορρίφθηκε η 80 υπέρ κατά απόχες εγκρίθηκε όχι διαμαρτυρίες. Εντάξει, ψηφίζουμε. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την 80. Άρχεται. Άρχεται η ψηφοφορία λοιπόν. Πέρας ψηφοφορίας. Ψηφίζουμε την 80. Πέρας ψηφοφορίας. 23 εναντίον 18 υπέρ απορρίφθηκε. Τώρα, οι τροπολογίες 81 και 82 είναι ταυτόσιμες. Ψηφίζουμε υπέρ αυτών. Κατά αποχές απορρίφθηκαν. Περνάμε στην προφορική τροποποίηση του εισηγητή στην παράγραφο 14. Έχουμε προφορική τροποποίηση, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. Η τροπολογία 83 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 84 υπέρ κατά αποχές Α, εγκρίθηκε, εγκρίθηκε μάλιστα η 84 και περνάμε στην Λίμπε 16 τροπολογία. Δύο τμήματα εδώ. Το πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Εγκρίθηκε, διορθώνει η πρόεδρος, εγκρίθηκε το πρώτο τμήμα. Εγκρίθηκε έτσι λοιπόν, μάλιστα εγκρίθηκε. Και το δεύτερο τμήμα τώρα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. ΦΑΜ 11 τροπολογία, υπέρ, γυναικών 11, υπέρ, κατά, νομίζω απορρίφθηκε. Και έτσι περνάμε στην τροπολογία 85 τώρα. Υπέρ. Α, την τροπολογία γυναικών, την 11, να την ελέγξουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την ΦΑΜ 11. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορία. 15 υπέρ, 27 εναντίον, απορρίφθηκε πράγματι. Τροπολογία 85 τώρα. Υπέρ. Υπέρ κατά άποχες απορρίφθηκε. Τροπολογία 86. Καταπίπτει αυτή. Επειδή εγκρίθηκε ο συμβιβασμός C. Και περνάμε στην Λίμπε 17. Υπέρ. Λίμπε 17. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Και περνάμε στην 87 τροπολογία. 87 υπέρ, κατά, αποχές απορρίφθηκε 88 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε φαμ 6 γυναικών 6 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε φαμ 9 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε περνάμε στην 89 τροπολογία υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 90 90 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 91 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε η 91 λίμπε 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε φαμ 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 92 τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 93 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε συμβιβασμός ή ε στη 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε και περνάμε στην τροπολογία 99 οι άλλες κατέπεσαν 99 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 100 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 101 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 102 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 103 υπέρ κατά 103. Τροπολογία 103. Παρακαλώ, ψηφίζουμε. Υπέρ. 103. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε η 103. 104. Υπέρ. Τροπολογία 104. Λοιπόν, υπάρχουν διαφορές στο ΕΛΚ. Θα ελέγξουμε γι' αυτό. Ε, είναι πολύ δύσκολο διαφορετικά να δει κανείς τι γίνεται. 104 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται. 104 τροπολογία. Πέρας ψηφοφορίας. Καταψηφίστηκε, απορρίφθηκε, ισοψηφία 21-21. Σαφής ο διαχωρισμός απορρίφθηκε λοιπόν. 21-21 ισοψηφία. ΦΑΜ 2 υπέρ. Τροπολογία ΦΑΜ 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. <clears throat> απορρίφθηκε. Η τροπολογία 105 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Εγκρίθηκε. Η 106 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Η 107 υπέρ κατά. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία, ψηφίζουμε την 107. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα εγκρίθηκε. 21 υπέρ, 18 εναντίον. Μια αποχή. Περνάμε στην παράγραφο 18. Συμβιβασμός F υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Περνάμε στην τροπολογία 111 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 112 τώρα υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Η 113 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Πάμε στην 114 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 115 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Περνάμε στην παράγραφο 20 συμβιβασμός G υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Περνάμε στην 118 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Η 119 τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Η 120 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Η 121 υπέρ κατά αποχές νομίζω εγκρίθηκε αλλά θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για να δούμε το αποτέλεσμα. Η 121 άρχεται. Άρχεται η ψηφοφορία, ψηφίζουμε την 121 πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα άλλη μια φορά ισοψηφία καταψηφίστηκε, απορρίφθηκε. Είχαμε ισοψηφία 21-21. 122 τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. Η 123 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. Η 124 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. ΦΑΜ 7, Επιτροπής Γυναικών 7, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. 125 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. 126 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. 127 υπέρ, κατά, αποχές απορρίφθηκε η 127. Η 128 υπέρ, κατά, αποχές απορρίφθηκε η 128. 129 υπέρ κατά άποχες εγκρίθηκε 131 καταπίπτει 131 γιατί εγκρίθηκε 129 το ίδιο ισχύει και για την 130 και περνάμε στην 132 τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 133 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά, αποχές εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, συγγνώμη, δεύτερο τμήμα και πάλι, της 133, δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίφθηκε το δεύτερο τμήμα. 134 τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Η 135 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. 136 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 137 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 138 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Περνάμε στην παράγραφο 24 συμβιβασμός H υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Πάμε στην στις άλλες τροπολογίες, στην παράγραφο 26, 142, 143, 144. Η 143 αποσύρθηκε, μάλιστα. Οι άλλες 2, 142, 144 είναι ταυτόσιμες, υπέρ αυτών, κατά αποχές. Απορρίφθηκαν οι 142, 144. Περνάμε στο συμβιβασμό I, υπέρ, κατά αποχές. Εγκρίθηκε. Περνάμε στην τροπολογία 149. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Η 150. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε η 150. Η 151. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω εγκρίθηκε. Περνάμε στην ΦΑΜ 8, Επιτροπής Γυναικών 8, υπέρ, κατά, <clears throat> αποχές, απορρίφθηκε. Περνάμε στην παράγραφο 28, συμβιβασμός J, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Λίμπε 2, τροπολογία, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. Πάμε στην 157 τροπολογία, υπέρ, κατά αποχές απορρίφθηκε η τροπολογία 6 τώρα υπέρ κατά απορρίφθηκε η 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε λίμπε α λίμπε α υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε λίμπε β λίμπε β υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Η τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Περνάμε στο αιτιολογικό β συμβιβασμός K υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Πάμε στην τροπολογία 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Περνάμε στην τροπολογία 15 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Η 16. Πώς είπατε. Τροπολογία 16 είπα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε Εγκρίθηκε, εγκρίθηκε διορθώνω. Τροπολογία 19 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. Τροπολογία 20 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Περνάμε στον συμβιβασμό L, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Περνάμε στην τροπολογία 23, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. Τροπολογία 24, υπέρ, κατά, αποχές απορρίφθηκε. Τροπολογία 25 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. Φαμ A, φαμ α, τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. Φαμ B, β, υπέρ, κατά, αποχές απορρίφθηκε. Φαμ C, γ, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. Λίμπε, σκεπτικό 1, υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. Λίμπε 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Πάμε στις τροπολογίες τώρα. 1 έως 6. Μπορούμε να τις ψηφίσουμε από κοινού. 1, 2, 3, 4 και 5 μέχρι την 6. Είναι κάποιος αντίθετος να ψηφίσουμε από κοινού όλες αυτές. Είσαστε αντίθετος. Μπορούμε να ψηφίσουμε λοιπόν από κοινού. Όλες μαζί. Ωραία. Να τις ψηφίσουμε 1, 2, 3, 4 και 5 από κοινού υπέρ αυτών, κατά, αποχές, εγκρίθηκαν, εγκρίθηκαν, σωστό, εγκρίθηκαν. Λίμπε τώρα, στο σκεπτικό 8, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Και η αιτιολογική σκέψη για, για το 10, λίμπε 4, η λίμπε 4 τροπολογία. Έχουμε την ΛΥΜΠΕ 4. Αιτιολογική σκέψη υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. Και τώρα, για την τελική ψηφοφορία ονομαστικά με ονομαστική κλίση, τελική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε στην τελική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας και αποτέλεσμα 37 υπέρ, 4 εναντίον, 3 αποχές. Εγκρίθηκε. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Και τώρα θα περάσουμε στη γνωμοδότηση της κυρίας Μπάουερ για την απορρόφηση των πόρων των διαθετικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής. Συναγόμενα διδάγματα για την πολιτική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. E então, eh, parágrafo primeiro... E- Πρώτη παράγραφος, τροπολογία 5, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. Περνάμε στον συμβιβασμό B υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Και περνάμε, οι άλλες καταπίπτουν, συμβιβασμό C γάμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Καταπίπτουν τα υπόλοιπα 11 θα την ψηφίσουμε ως ε, αιτιολογική σκέψη υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε η 12 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε η 13 υπέρ, κατά, αποχές απορρίφθηκε 14 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε 15 υπέρ κατά αποχές δεν είμαι βέβαιη για το αποτέλεσμα καλύτερα να ελέγξουμε ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 15 άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας 21 a 22 κόντρα. 21 υπέρ 22 εναντίον απορρίφθηκε η 16 καταπίπτει επειδή εγκρίθηκε ο συμβιβασμός περνάμε στον συμβιβασμό D υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε και περνάμε στην 21 οι άλλες καταπίπτουν υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 22 αποσύρθηκε. Περνάμε στον συμβιβασμό Ή υπέρ. Κατά αποχέσα εγκρίθηκε. Και περνάμε έτσι στην 29. Γιατί εντωμεταξύ... Α, εντάξει, η 23 είναι συμβατή με τις προηγούμενες τροπολογίες. Και γι' αυτό λοιπόν θα ψηφίσουμε την 23 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Το ίδιο και για την 24 υπέρ κατά αποχές. Νομίζω απορρίφθηκε. 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 29 υπέρ κατά αποχές Δεν είμαι καθόλου βέβαιη αν απορρίφθηκε ή όχι. Προτιμώ να υπαλληθεύσουμε. Ψηφίζουμε την 29. Άρχεται η ψηφοφορία. 29 τροπολογία. Ε, Πέρας ψηφοφορίας. Απερίφθη μάλιστα. Απορρίφθηκε. Ζητώ συγγνώμη. Η 31 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Συμβιβασμός F. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Περνάμε στον συμβιβασμό G. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Περνάμε στην τροπολογία 33. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Τροπολογία 34. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Τροπολογία 35. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίφθηκε. Συμφασμός H υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Και περνάμε τώρα στην τροπολογία 40 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Συμβιβασμός E, I, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Και περνάμε στην τροπολογία 42 υπέρ κατά αποχές απο... εγκρίθηκε η ορθόνη πρόεδρος εγκρίθηκε η 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε η 45 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε συμβιβασμός J υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε πάμε στον συμβιβασμό K υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Και περνάμε στην τροπολογία 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 55 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 56 καταπίπτει η 56 και περνάμε στην 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε συμβασμός ε, L υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 64 τροπολογία υπέρ κατά αποχές Απορρίφθηκε η 64. Η 65. Να ελέγξουμε την 64. Ελέγχουμε την 64. Ψηφίζουμε άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας και αποτέλεσμα απορρίφθηκε. 20 υπέρ 21 εναντίον. Απορρίφθηκε. Και τώρα τροπολογία 65 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός Α, Α υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Και τελική ψηφοφορία τώρα Άρχεται η ψηφοφορία και τώρα πέρας ψηφοφορίας. 42 ψηφίσαντες, 39 υπέρ, ενα εναντίον, δύο αποχές. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια, στην κυρία Μπάουερ. Και έτσι ολοκληρώσαμε τις ψηφοφορίες, αυτή την ψηφοφορία και θα περάσουμε στην επόμενη όπου έχουμε και εδώ μια γνωμοδότηση του κυρίου Dirk Sterks, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κίνα, μια εμπορική ανισορροπία. Συγητής ο κύριος συντάξει γνωμοδότηση ο κύριος Dirk Sterks. Περνάμε στην ψηφοφορία. Τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Συμβιβασμός C γάμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Περνάμε στην τροπολογία 6. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. Συμβιβασμός A, α, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Τροπολογία 8 όχι, τροπολογία 8 καταπίπτει, μάλιστα, και αυτή καταπίπτει. Και η 9 καταπίπτει. Η 10, η 11, 12 καταπίπτουν όλες, φτάνουμε στη 14. Τροπολογία 14 λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίθηκε. 15 υπέρ. Κατά. Απόχες. Απορρίφθηκε. 16 υπέρ. Κατά. Απόχες. Απορρίφθηκε. 17 υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. 18 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Εν τω μεταξύ 19 αποσύρθηκε, 20 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 20. Περνάμε στον συμβιβασμό Β, Β υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Πάμε τώρα στην τροπολογία 23, 22 δεν ήταν αποδεκτή. 23 και 24 έχουν ήδη καλυφθεί και 25 και αυτοί. Περνάμε στο συμβιβασμό D, δέλτα. Συμβιβασμός D, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Περνάμε τώρα στη συνέχεια στην τροπολογία 29. Οι άλλες κατέπεσαν 27 και 28. 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 30 Συγγνώμη, συγγνώμη, 29. 29 νομίζω εγκρίθηκε, αλλά υπάρχει αμφιβολία και πρέπει να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία στην 29. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 27 υπέρ 14 εναντίον, σαφές το αποτέλεσμα εγκρίθηκε, υπεψηφίστηκε. Η 30 τροπολογία, υπέρ. κατά αποχές απορρίφθηκε 31 διαμαρτυρία 31 και 32 κατέπεσαν πάμε στην 33 με προφορική τροποποίηση του κυρίου Χέλμερ. υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 34 υπέρ κατά Δεν είναι σαφέ το αποτέλεσμα. Ζητώ συγγνώμη. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά γιατί δεν ήταν σαφέ το αποτέλεσμα. Άρχεται η ψηφοφορία. 34. Πέρας ψηφοφορία τώρα. 31 υπέρ 10 εναντίον. Εγκρίθηκε. 35. Πρώτο τμήμα γιατί το δεύτερο δεν είναι αποδεκτό σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη. Ψήφι υπέρ του πρώτου τμήματος κατά αποχές εγκρίθηκε το πρώτο τμήμα. Και πάμε στην τροπολογία 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 38 υπέρ κατά αποχές Απορρίφθηκε η 38. 39. Κατέπεσε η 39. Μια και εγκρίθηκε ο συμβιβασμός. Περνάμε στη 40. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 41. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 42. Υπέρ Α, και αυτή κατέπεσε η 42. 42, 43, 44 κατέπεσαν. Περνάμε στην 45, 46. Είναι ταυτόσιμες οι δύο αυτές. Υπέρ αυτών, κατά, αποχές, απορρίφθηκαν. 47, 47, ψηφίσουμε γιατί δεν εγκρίθηκαν οι προηγούμενες υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε η 47. 48 υπέρ, κατά, απόχες εγκρίθηκε 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 50 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε η 50 51 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε δεύτερο τμήμα δεν αξίζει να ψηφιστεί γιατί ούτως ή άλλως απορρίφθηκε το πρώτο Δεύτερο, έστω, υπέρ. Ωραία. Κατά, απόχες, απορρίφθηκε. Πάει και αυτό. Τροπολογία 52 της κυρίας Λάμπερτ, σε δύο τμήματα και αυτή. Πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά, απόχες. Καλύτερα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά, να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για το πρώτο τμήμα της 52. Πέρας ψηφοφορίας και αποτέλεσμα εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα τώρα της τροπολογίας αυτής υπέρ, κατά, αποχές. Το δεύτερο απορρίφθηκε όμως το δεύτερο τμήμα της. Καταπίπτουν οι δύο ακόλουθες τροπολογίες και φτάνουμε θα ψηφίσουμε την 55. Εντάξει, υπέρ. 55 υπέρ. Υπέρ. 55 κατά. Κατά. Απόχες. Νομίζω απορρίφθηκε. Αλλά να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Έτσι άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε την 55. Aberta a 55. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα εγκρίθηκε. Η 56 με προφορική τροποποίηση υπέρ κατά αποχές. Απορρίφθηκε. 57 υπέρ κατά αποχές. Απορρίφθηκε. 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 60. Τροπολογία 60. Γιατί η άλλη η 59 κατέπεσε. 60 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Νομίζω εγκρίθηκε έτσι. Ωραία. Περνάμε στην τροπολογία 1. Να ελέγξουμε την 60. Ωραία. Εγώ νομίζω ότι εγκρίθηκε, αλλά θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται. Ψηφίζουμε την 60. Το Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας λοιπόν. Και αποτέλεσμα εγκρίθηκε μάλιστα. Λοιπόν, 26 υπέρ, 17 εναντίον εγκρίθηκε. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. Τροπολογία 1. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά λοιπόν, θα ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε την τροπολογία 1 you Eu não me é mais um bocado ou menos 12. Απορρίφθηκε 12 υπέρ, 28 εναντίον. Απορρίφθηκε. Η τροπολογία 2 τώρα υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίθηκε η 2. Τροπολογία 3 υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίφθηκε, απορρίφθηκε η τρία. Και τώρα πάμε στην τελική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά, τελική ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας, ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 35 υπέρ, 6 εναντίον και 2 αποχές. Συγχαρητήρια στον εισηγητή μας. Εγκρίθηκε η γνωμοδότηση. Ε, Και τώρα μπορούμε... Ε, Εδώ, παρότι έχουμε την ένδειξη ότι έχουμε ένα θέμα, προφορικό αίτημα, για τη διανομή τροφίμων, αυτή η ερώτηση αντικαταστάθηκε από μια προφορική ερώτηση για τους άστεγους. Για τους άστεγους, για προφορική ερώτηση για τους άστεγους. Τίθεται σε ψήφιση λοιπόν, σε ψηφοφορία. Στη συνεδρία των συντονιστών εγκρίθηκε αυτή η αντικατάσταση με μια προφορική ερώτηση και με ένα ψήφισμα που θα ακολουθεί την προφορική ερώτηση. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά να δούμε αν εγκρίνουμε. Πρώτα την προφορική ερώτηση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ε, Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 37 υπέρ 5 εναντίον. Υπερψηφίστηκε, εγκρίθηκε. Και μετά έχουμε και το δεύτερο θέμα. Δεύτερη ψηφοφορία για το ψήφισμα. Πρόταση ψηφίσματο. Άρχεται η ψηφοφορία. Eh, Ψηφίζουμε, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας τώρα. Και αποτέλεσμα. 38 υπέρ, 5 εναντίον εγκρίθηκε η κατάθεση ψηφίσματος. Και ολοκληρώσαμε λοιπόν εδώ την περίοδο ψηφοφοριών, τις ψηφοφορίες μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλες και όλους σας για τη συνεργασία σας σε αυτές τις ψηφοφορίες. Σε αυτή τη συνεδρίαση που είχαμε κάποιες περιπλοκές. Ο συνάδελφός μας, Ρώσα, ζήτησε τον λόγο. Έχετε τον λόγο. Uh, uh, επανέλθουμε στην ημερήσια διάταξη. Ε, Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μου δίνει η γραμματεία, παρούσα στην διάσκεψη προέδρων. η Πρόεδρη θα είναι εκείνη, Η διάσκεψη των προέδρων θα αποφασίσει αυτή την ερώτηση. Αν θα κατατεθεί ή όχι στην Ολομέλεια η ερώτηση αυτή. Σε ευχαριστώ. Então, depois do Λοιπόν, μετά από την περίοδο αυτή που είχαμε τις ψηφοφορίες, θα περάσουμε τώρα με μια μικρή, μικρή, πολύ μικρή καθυστέρηση στη συζήτηση του σημείου 19 στην ημερήσια διάταξη. Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας, καταπολέμηση της φτώχειας και του, κοινωνικού αποκλεισμού. Η συγητής μας είναι ο κύριος Φρεντερίκ Νταρντόν. Του δίνω αμέσως τον λόγο. Έχετε τον λόγο κύριε Νταρντόν για να μας παρουσιάσετε το σχέδιο έκθεσή σας και για τις απόψεις που έχετε να μας παρουσιάσετε και θα αρχίσουμε τη συζήτηση μετά. Έχετε τον λόγο κύριε αγαπητέ συνάδελφε Νταρντόν. Ζητώ όλοι οι άλλοι συνάδελφοι παρακαλώ <clears throat> και από τη γραμματεία επίσης να καθίσουν στις θέσεις τους και να είναι ήσυχοι παρακαλώ, ησυχία ώστε ο συνάδελφός μας να μπορεί να μας προσφωνήσει όπως πρέπει μέσα σε ένα περιβάλλον ησυχίας, ηρεμίας. Ε, Παρακαλώ και πάλι η γραμματεία όσοι και όσοι βουλευτές ε, βρίσκονται εδώ να καθίσουν να καθίσετε όλοι στις θέσεις σας. Έχετε τον λόγο κύριε αγαπητέ συνάδελφε Φρέντερικ Ντάντον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί φίλοι, υπάρχουν μερικά, μερικές γενικές παρατηρήσεις προτού ασχοληθώ με το περιεχόμενο της έκθεσης. Η έκθεση εντάσσεται μέσα στην, στο πλαίσιο της στρατηγικής 2020 που προβλέπει μείωση 20 εκατομμυρίων ατόμων που βρίσκονται σε επισφαλή κατάσταση. Δεν ξέρω αν αυτή η μείωση είναι επαρκής ή αν δεν είναι αρκετά φιλόδοξη. Δεν είναι αυτό το αντικείμενο αυτής της έκθεσης. Νομίζω ότι ο στόχος είναι τώρα να μπορέσουμε το 2020 να επιτύχουμε 20 εκατομμύρια άτομα να βγουν από την επισφαλή κατάσταση. Πρόκειται από τις σημαντικές εμβληματικές ε, πρωτοβουλίες και εντάσσεται στην πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας της Κομισιόν. Συμφωνούμε όλοι ότι η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός που δυστυχώς αυξάνουν χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Προκύπτει από τις διάφορες συζητήσεις ότι αυτή η φτώχεια έχει πολλές πηγές, πολλές απόψεις, πολλά σκέλη ε, και θίγει τα παιδιά, τους υπερήλικες, ε, τους ανάπηρους, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, τους μετανάστες, αυτούς πλήττει και υπάρχει σχέση ανάμεσα στη φτώχεια και στην καταπολέμηση της φτώχειας και στον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αν ορισμένοι διατείνονται ότι η καταπολέμηση της φτώχειας είναι ουσιαστικά της αρμοδιότητας, των κρατών, εμένα μου φαίνεται αναμφισβήτητο ότι η Ευρώπη έχει ένα ρόλο να παίξει στον τομέα αυτών Εξάλλου, κατά τη διάρκεια του 2010, του περσίνου έτους, στο πλαίσιο της εκπόνησης της στρατηγικής 2020 και στα πλαίσιο του έτους καταπολέμησης της φτώχειας, πάρα πολλά σε πολλές συζητήσεις, πολλά επιχειρήματα υποβλήθηκαν κυρίως μέσα σε αυτό το κοινοβούλιο. Εκπώνησα λοιπόν αυτό το σχέδιο εισήγησης ξεκινώντας από τις, τους συλλογισμούς αυτούς και από τις συζητήσεις που άπτονται κλασικών θεμάτων της Επιτροπής μας. Εκπώνησα επίσης αυτό το σχέδιο έκθεσης βάσει των επαφών που είχαμε πάρα πολλές οργανώσεις που ασχολούνται με τον τομέα αυτό και νομίζω ότι μερικές εκπροσωπούνται σήμερα εδώ, στην αίθουσά μας. Θα ήθελα τώρα ε, να αναφερθώ στο περιεχόμενο του σχεδίου εισήγησης πέραν από ε, τα εκτιμώντας από την αιτιολογική έκθεση υπάρχουν μερικές ε, προτάσεις ως προς τη μέθοδο και τις ε, γενικές αρχές. Επαναλαμβάνουμε εδώ την αναγκαιότητα της συμμετοχής στα πλαίσια της πλατφόρμας των οργανώσεων και των ατόμων που βρίσκονται σε επισφαλή κατάσταση. Επιμένουμε επίσης πάνω στην ανάγκη της υλοποίησης ε, της οριζόντιας κοινωνικής διάταξης, την ενίσχυση του συντονισμού στον κοινωνικό τομέα την απαραίτητη ενσωμάτωση στον προϋπολογισμό των ευρωπαϊκών δράσεων σε σχέση με την καταπολέμηση της φτώχειας αλλά και ενσωμάτωση στους προϋπολογισμούς των κρατών και πρέπει να αφήσουμε στα κράτη περιθώρια δημοσιονομικά κυρίως στα πλαίσια της επίκαιρης συζήτηση της οικονομικής διακυβέρνησης πρέπει λοιπόν να υπάρξουν περιθώρια ε, δαπανών που ευνοούν την απασχόληση, την κοινωνική ενσωμάτωση. Αν μειωθούν οι κοινωνικές διαπάνες, αυτό θα έρχεται σε αντίθεση με τον στόχο της μείωσης της φτώχειας. Πρέπει επίσης να ελέγξουμε τις προσπάθειες που καταβάλλονται από τα κράτη-μέλη, κυρίως για την υλοποίηση των συστάσεων σχετικά με τα μέτρα συμπερίληψης ενσωμάτωσης. Πρέπει επίσης να ευνοήσουμε ένα ολόκληρο φάσμα δικτών ευρωπαϊκών για την μέτρηση της φτώχειας, όχι μόνο το κατόφλι της φτώχειας, αλλά θα πρέπει να διευκρινίσουμε καλύτερα τα προβλήματα, την εξέλιξη της φτώχειας για κάθε κράτος ε, και κάθε στάδιο. Θα πρέπει επίσης να υπάρξει μια παρακολούθηση τακτική με συμμετοχή του Κοινοβουλίου για την υλοποίηση αυτές της πλατφόρμας. Πέραν των προτάσεων αυτών των προτάσεων αυτών για τη μέθοδο και τις γενικές αρχές. Μερικά θέματα πιο ειδικά αναφέρονται. Ο ρόλος του ελάχιστου εισοδήματος έγινε ήδη λόγος γι' αυτό κυρία Πρόεδρε, ο ρόλος της κατάρτισης, της εκπαίδευσης, ο ρόλος των κοινωνικών υπηρεσιών κοινή ωφέλεια, επίσης οι επιπτώσεις της στέγης, της κατοικίας, της ενέργειας, στην φτώχεια, ο ρόλος των διαφορετικών ταμείων ε, για να βγουν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες από τη φτώχεια. Αυτά τα θέματα αναφέρονται στην εισήγηση αυτή. Είναι προφανές ότι η εισήγηση αυτή θα πρέπει να συμπληρωθεί, να διευκρινιστεί, να προσδιοριστεί καλύτερα, αλλά χρειάστηκε ε, λόγω έλλειψης ε, χώρου, χρόνου, ε, να κάνουμε την αυτοκριτική μας, την αυτολογοκρισία μας κατά κάποιο τρόπο και έχουμε ήδη μια σειρά τροπολογιών που είναι έτοιμες για κατάθεση για να συμπληρωθεί αυτό το κείμενο. Υπάρχουν επίσης και οι γνωμοδοτήσεις στις επιτροπές που θα έρθουν να συμπληρώσουν την έκθεση. Έχουμε την Επιτροπή Προϋπολογισμού, Επιτροπή Πολιτισμού, Επιτροπή Γυναικών. Όλα αυτά θα συμπληρώσουν την έκθεση. Είμαι πεπισμένος γι' αυτό και Σκέφτομαι επίσης ότι με τις τροπολογίες ε, και τις πρόσθετες ιδέες που θα μπορούσαν ε, να προσθεθούν ε, ή να διευκρινιστούν σε σχέση με τους άστεγους, την φτώχεια των παιδιών, τις συντάξεις. Αυτά είναι μερικά στοιχεία εισαγωγικά για την παρουσίαση της έκθεσής μου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Νταρντένα. Ήδη έχω έναν κατάλογο από σκιώδεις εισηγητές και από συναδέλφους που επιθυμούν να παρέμβουν και εγώ ίδια θα ήθελα να πω τα Η έκθεση η οποία εξετάζει ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Εξάλλου η Επιτροπή μας πέρσι απόδωσε μεγάλη σημασία στο θέμα αυτό στην έκθεση «Η Ευρώπη και η καταπολέμηση της φτώχειας». Εξάλλου κάναμε πολλές συστάσεις, θυμάμαι την έκθεση για την οποία είχα και εγώ εργαστεί πολύ για το ελάχιστο εισόδημα. Εν τω μεταξύ, έχουμε μια επιδίνωση της φτώχειας, της φτώχειας μεταξύ των οικογενειών και μεταξύ των παιδιών σε όλα τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη μας τα οποία αντιμετωπίζουν πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα σήμερα. Ο συνάδελφος επισύρει την προσοχή μας πάνω σε πάρα πολλές απόψεις και υπάρχουν και πολλές τροπολογίες. Εγώ θα επιθυμούσα να περιλάβουμε και άλλες απόψεις, άλλα σκέλη, δηλαδή τα αίτια της κατάστασης, τα μέτρα πιο δραστήριας πολιτικής με μεγαλύτερη αλληλεγγύη, μια πολιτική συνοχής οικονομικής και κοινωνικής, μια παρέμβαση, ε, μια δραστηριοποίηση μεγαλύτερη στο επίπεδο των κοινοτικών ταμείων. Αυτή είναι μια ολόκληρη σειρά ιδεών που προτάσω ως κοιόδης εισηγήτρια της ομάδας μας για τροπολογίες που ασφαλώς θα παρουσιάσουμε για την έκθεσή σας. Και δίνω αμέσως το λόγο το, στον κύριο Λόπ Φοντανιέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω στον εισηγητή ότι άκουσα πολύ καλά ότι μας είπε ότι πρόκειται να παρουσιάσει και άλλες τροπολογίες. Δεν μπόρεσε να περιλάβει όλες αυτές τις τροπολογίες στην έκθεσή του, να τις εντάξει. Αλλά εγώ θα έλεγα ότι αυτό είναι κάτι το πάρα πολύ συγκεκριμένο. Καλύπτει όλα τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας και είμαι βέβαιη ότι με τον εισηγητή θα μπορέσουμε να παρουσιάσουμε μια εισήγηση που θα καλύπτει όλα τα θέματα τα οποία δυστυχώς είναι θέματα μεγάλης επικαιρότητα λόγω της κρίσεως την οποία βιώνουμε. Νομίζω ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο. Θα πρέπει να μιλήσουμε για την πλατφόρμα γνωρίζοντας ότι ένα μεγάλο μέρος του προβλήματος εξαρτάται από τη βούληση των κρατών μελών. Νομίζω όμως ότι είναι μια εργασία πάρα πολύ σημαντική. Θα έχουμε τη δυνατότητα και το χρόνο να συζητήσουμε τις τροπολογίες, αλλά θα ήθελα να προτάξω διάφορα στοιχεία. Μίλησε για αυτό ο εισηγητής στις οικογένειες ή στα παιδιά. Εγώ δεν θα μιλούσα πάντοτε για οικογένειες. Όλα εξαρτώνται βεβαίως για τα παιδιά από τη φτώχεια των οικογενειών, τα υπερήλικες και τα εξαρτώμενα άτομα. δεν είναι επειδή είναι εξαρτώμενα, επειδή είναι υπερήλικες που βρίσκονται σε επισφαλή κατάσταση. Αυτό σχετίζεται με την εγκατάλειψη, την μοναξιά, τον κοινωνικό αποκλεισμό. Θα πρέπει να συγκεντρωθούμε πάνω στα θέματα αυτά, κυρίως όσον αφορά στις γυναίκες. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να υποβάλουμε πολλές τροπολογίες για τις γυναίκες, εφόσον υπάρχει ήδη μια έκθεση, μάλλον μια γνωμοδότηση για τις γυναίκες. Αλλά εγώ δεν αποκλείω τις γυναίκες που είναι μόνες τους, που έχουν, επιβαρύνονται με παιδιά ε, και για τους Αθήγανους. Νομίζω ότι για μας είναι σημαντικό είναι σημαντικό αυτό, ε, αυτές οι ομάδες να περιληφθούν παντού στην πλατφόρμα. Δεν πρέπει να ξεχνούμε επίσης τις οργανώσεις, τις κοινωνικές που εργάζονται με τους Ρωμά εδώ και χρόνια και που έχουν βεβαίως πολλά να πούν και πολλά να προσφέρουν για να αναπτύξουμε καλά την συμπερίληψη των ευπαθών αυτών ατόμων. Ο εισηγητής μας είπε ότι υπάρχουν δύο σημεία στα οποία θα διορθώσει την σύνταξη, την οδηγία, την οριζόντια για τον αποκλεισμό. Αυτό δεν ξέρω αν περιλαμβάνεται στην συνθήκη, μπορούμε πάντοτε ε, να δώσουμε μια νέα τροπή στο κείμενο για την οδηγία και το άρθρο 18, η οδηγία πλαίσιο για τον ελάχιστο μισθό. Τον... Υπάρχουν πάρα πολύ καλές ιδέες, αλλά δεν ξέρω τι θα γίνει. Η πρόεδρος έκανε μια έκθεση για το θέμα αυτό, αλλά είναι δύσκολο να εναρμονιστούν τα συστήματα ε, κοινωνικής προστασίας όλων των κρατών μελών. Θα πρέπει ε, να ασχοληθούμε εντατικά με το θέμα αυτό ε, που είναι ένα θέμα σημαντικό αλλά το οποίο έχει πολλά περίπλοκα σημεία. Εξ ονόματος της ομάδας μου είμαστε στη διάθεσή σας κυρία Πρόεδρε για να εργαστούμε και να παρουσιάσουμε τροπολογίες οι οποίες θα μπορέσουν να είναι χρήσιμες για την έκθεσή σας. E Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Λίνα έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστούμε κυρία Λίνα. Βεβαίως υπάρχουν ε, πολύ θετικά στοιχεία ε, στην ε, γνωμοδότηση στο G συμφωνείτε, αλλά εμείς χρησιμοποιούμε άλλους δείκτες ε, φτώχειας. Νομίζω λοιπόν ότι ίσως καλό θα ήταν να το δούμε γιατί δεν υπάρχει ένας δείκτης ε, ένδυας ε, που χρησιμοποιείται παντού. Σχετικά με το 10. Θέλουμε ε, στο 10 να αναφέρουμε ε, την οδηγία για την ε, απασχόληση, τα μέτρα τα οποία αφορούν την εξέβρεση εργασίας. Νομίζω ότι θα πρέπει να το δούμε αυτό. Και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για, τους, για τα άτομα με αναπηρία. 13. Λοιπόν, η Επιτροπή έχει ήδη ξεκινήσει μια οδηγία κατά των ε, διακρίσεων που έχει φτάσει ε, στην, ε, στο Συμβούλιο και επομένως νομίζω ότι θα πρέπει να αλλάξει λίγο η διατύπωση. Ε, όχι ζητά να υπάρξει οριζόντια οδηγία γιατί υπάρχει πλέον, υφίσταται η οριζόντια αυτή οδηγία κατά των διακρίσεων. 18. Α, να πω και κάτι άλλο. Κάτι που ανέφερε και η κυρία Φιγκερέιδα. Ε, νομίζω ότι και στην προηγούμενη έκθεση της κυρία, που συνέταξε η κυρία Φιγκερέιδα. Ε, θα, ότι πρέπει να πούμε ε, τι εννοούμε όταν αναφέρουμε ελάχιστο μισθό και ελάχιστη αμοιβή. Ο ελάχιστος μισθός ε, είναι αυτός που καθορίζουν οι κοινωνικοί εταίροι ή η νομοθεσία στα κράτη-μέλη όσον αφορά την απασχόληση. Αυτός είναι ο ελάχιστος μισθός. Το ελάχιστο εισόδημα όμως ε, είναι το εισόδημα το οποίο έχουν άνθρωποι οι οποίοι συνήθως δεν εργάζονται μέσω επιδομάτων κοινωνικής ασφάλισης κτλ. Ε, κάποιοι πολύ χαμηλόμιστοι εργαζόμενοι ίσως χρειαστούν και το ελάχιστο εισόδημα. Πάντως όταν μιλάμε για ελάχιστο εισόδημα αναφερόμαστε στο ε, ελάχιστο ποσοστό το οποίο χρειάζεται στις διάφορες χώρες μέλη για την επιβίωση. Ενώ η ελάχιστη αμοιβή, ο ελάχιστος μισθός είναι κάτι διαφορετικό. Ας πούμε, εσείς αναφέρεστε σε συλλογικές διαπραγματεύσεις ε, για ελάχιστο κειμένο εισόδημα. Προφανώς όμως θα πρέπει να αναφέρετε το ελάχιστο, ε, ε, τον ελάχιστο κειμένο μισθό, γιατί το εισόδημα είναι τελείως διαφορετικό. Ε, εγγυημένο εισόδημα συνήθως αναφέρεται σε ανθρώπους που δεν βρίσκονται ε, στην αγορά εργασίας, δηλαδή δεν έχουν απασχόληση, είναι στην ανεργία ή δεν μπορούν να εργαστούν ε, νομίζω ότι αυτό το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα ε, είναι λίγο διαφορετικό πράγμα. Ξέρω ότι γίνεται λόγος τώρα για ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα που θα λαμβάνουν κάποιοι άνθρωποι, αλλά ε, σε ανταπόδοση θα κάνουν κάποια κοινωνική εργασία ή κάτι τέτοιο. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε οδηγία πλαίσιο σχετικά με το ελάχιστο εισόδημα. Γιατί αυτό που βλέπουμε στα κράτη-μέλη και μετά από τα νέα κράτη-μέλη είναι ότι έχουν πρόβλημα και εν πάση περιπτώσει αντιμετωπίζουν με τρόπο τελείως διαφορετικό το θέμα του εισοδήματος. Νομίζω λοιπόν ότι είναι εσφαλμένο σε αυτή τη χρονική στιγμή να μιλήσουμε για οδηγία πλαίσιο ε, για ελάχιστο κείμενο εισόδημα, αλλά βεβαίως ε, ε, σε βασμό των πρακτικών, ναι, φυσικά. Στο 19 αναφέρεται τα ηλικιωμένα άτομα. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Οπότε μιλάμε ε, όταν μιλάμε για ηλικιωμένα άτομα ε, ε Ε, στα αγγλικά ε, δεν λέμε ποτέ ηλικιωμένοι ή ανάπηροι, λέμε ηλικιωμένα άτομα, ηλικιωμένοι άνθρωποι κτλ. Ε, λοιπόν, όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά που λέτε να αναπτυχθούν συστήματα αμέριμνας, ε, και να αποτραπεί το γεγονός να βρεθούν οι άνθρωποι αυτοί σε κατάσταση κοινωνικού αποκλεισμού ή φτώχειας. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα των ηλικιωμένων γενικότερα ε, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν δηλαδή οι ηλικιωμένοι ε, όσον αφορά τη φτώχεια, όσον αφορά τον κοινωνικό αποκλεισμό κτλ. Δηλαδή κατά κάποιο τρόπο πιο εμφατικά να αναφερθούμε στα σημεία αυτά. Ευχαριστώ πολύ λέει η Πρόεδρος. Πάρα πολύ ωραία. Πριν προχωρήσουμε, νομίζω ότι θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε δύο πράγματα, να αποσαφηνίσουμε. Πρώτον, η έκθεσή μου αφορούσε αφορούσε το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Ε, ελάχιστο εισόδημα και εγώ δεν ενέφερα καθόλου το θέμα του ελάχιστου μισθού. Ελάχιστο εισόδημα, δηλαδή μέσω κοινωνικών επιδομάτων που θα πρέπει να δοθούν σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τα μέσα για να επιβιώσουν. Εμείς ε, πέρσι είχαμε ζητήσει λοιπόν αυτό το εγγυημένο εισόδημα που πρέπει να είναι το 60% του ε, μισθού ε, στις, ε, σε κάθε χώρα, όχι του ευρωπαϊκού μεσόρου, με, αλλά σε σχέση με τα ισχύοντα σε κάθε χώρα. Εμείς ορίσαμε το 60%, 60 του εισοδήματος της κάθε χώρας, έτσι ώστε για κάθε χώρα το ποσό να είναι διαφορετικό. Δεν πρέπει να μπερδεύουμε λοιπόν το εισόδημα με το μισθό, το ελάχιστο εισόδημα με τον ελάχιστο μισθό. Έστω και αν προτείνουμε βεβαίως να υπάρχει ένας ελάχιστος μισθός σε κάθε χώρα, ε, λαμβάνοντας υπόψη φυσικά τις συλλογικές συμβάσεις, συλλογικές διαπραγματεύσεις, ε, τα είδη των ε, συμβάσεων που υπάρχουν σε κάθε χώρα κτλ. Και πάντα επόμενη την αρχή της επικουρικότητας φυσικά. μερικές φορές δεν γίνεται διαχωρισμός ανάμεσα στο εισόδημα και το μισθό, αλλά πρέπει να είμαστε σαφείς. Η έκθεσή μου αναφερόταν στην, ε, στον ελάχιστο, στο ελάχιστο εισόδημα και όχι στον ελάχιστο μισθό. Αυτά. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Κουζαλόφσκι, τον συνάδελφό μας. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ως σκιώδης από την πλευρά της Επιτροπής των Προϋπολογισμών θα ήθελα να πω και εγώ δύο λόγια και να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις. Πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τον Σνάρφο Ντερντέν γιατί η έκθεσή του αναφέρεται σε πολλά και σημαντικά θέματα είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τη δικιά μας Επιτροπή εδώ, αλλά και για την Επιτροπή Προϋπολογισμών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει αναλυτική χρήση, ε, αναλυτική συγγνώμη παρουσίαση των ε, κονδυλίων για την πλατφόρμα για την φτώχεια ε, και τα λοιπά. Εγώ όμως δεν θα συμφωνήσω με τα όσα αναφέρεται ε, στο σημείο 9 ζητά ισότητα των δικαιωμάτων και κοινωνικής προστασίας για όλους τους εργαζόμενους σε κάθε κράτες μέλους. Γιατί εδώ μπαίνουμε στα χωράφια του κράτους ε, μέλους. Δηλαδή υπάρχουν και εθνικές προτεραιότητες και ιδιαιτερότητες. Πάντως συμφωνώ με την παρουσίαση που κάνει ο συνάδελφος Νταρντέν για τις ε, ομάδες ε, οι οποίες αντιμετωπίζουν φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό. Και να σας πω ότι στις 17 ε, και 18 Οκτωβρίου 2011 στην Κρακοβία, θα, στην Πολωνία δηλαδή, υπό Πολωνική Προεδρία, θα, πρε, θα λάβει χώρα η πρώτη συνάντηση της ε, πλατφόρμας και πιστεύω ότι όλα αυτά τα θέματα ε, θα τα συζητήσουμε. Επίσης ε, είναι παράδεκτο να μιλάμε για γυναίκες οι οποίες πέραν του ότι είναι γυναίκες, είναι άνεργες, έχουν στην φύλαξή τους παιδιά και αυτό είναι πραγματικά μεγάλη έκθεση στην φτώχεια. Ελπίζω επίσης το 2012, το οποίο έχει ε, οριστεί σαν ε, έτος της ενεργητικής ε, μεγάλης ηλικίας θα επιβεβαιώσει κάποια στοιχεία τα οποία ζητάει και ο κύριος Δερντένας όσον αφορά τους ηλικιωμένους. Επίσης ε, πιστεύω ότι όταν μιλάμε για άτομα με αναπηρία ε, θα πρέπει να τους λάβουμε ειδικά υπόψη μας. Πρέπει επίσης να πούμε ότι η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν αναφέρεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όμως τρία τέταρτα των θέσεων εργασίας στην Ευρώπη ε, στην ουσία προσφέρεται μέσω των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επομένως θα πρέπει να βοηθηθούν και η, ε, ο ρόλος τους μάλλον στην καταπολέμηση της ένδυας είναι πάρα πολύ μεγάλος. Ευχαριστώ. Η κυρία Νταλή. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Εισηγητά, αγαπητοί συνάδελφοι, εάν δεν μας αφήνετε να ονειρευόμαστε, εμείς δεν θα σας αφήσουμε να κοιμηθείτε. Οι νέοι οργισμένοι της Πουέρτα del Sol στη Μαδρίτη ανέφεραν με τα λόγια αυτά, εξέφρασαν την απόγνωσή τους απέναντι σε μια πολιτική τάξη που δεν μπορεί να φέρει συγκεκριμένες αυτές λύσεις ε, στα άτομα τα οποία υποφέρουν από τις τρομερές συνέπειες της κρίσης της πολιτικής, οικονομικής, περιβαλλοντικής και δημοκρατικές που ζούμε. Περίπου 23 εκατομμύρια άνεργοι στην Ευρώπη, πάνω από 85 εκατομμύρια άτομα που ζουν κάτω από το κατόφλι της φτώχειας, 116 εκατομμύρια άτομα που απειλούνται από τη φτώχεια. Οι νέοι πλήττονται δύο φορές περισσότερο από τον υπόλοιπο πληθυσμό από τους ανέργους. Ένας στους πέντε νέους ε, ζει στην φτώχεια, η απασχόληση ε, δεν ε, προστατεύει από την ένδια λόγω των επισφαλών συνθήκων εργασίας έχουμε τόσους Ευρωπαίους φτωχούς ενώ εργάζονται, απασχολούνται. Πώς μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι με αυτές τις διαπιστώσεις αυτή η κατάσταση είναι παραπάνω από απαράδεκτη. Γι' αυτό η εμβληματική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Καταπολέμησης της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού είναι μια πρωτοβουλία για να προχωρήσει αυτή η κοινωνική Ευρώπη υπέρ ε, των ε, πιο εσφαλών ε, και απόρων ε, Ευρωπαίων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Νταρντέν ε, για το σχέδιο έκθεσης, αλλά θα ήθελα να πω σε όλους ότι έχουμε ακόμα πάρα πολλά να κάνουμε και δεν έχουμε το δικαίωμα να αποτύχουμε το Ευρωπαϊκό Έτος Καταπολέμησης της Φτώχειας. Τι έχει αφήσει ως κληρονομιά. Τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Όλα απομένουν να γίνουν απορρίπτοντας την πρόταση μιας οδηγίας πλαισίου για το ελάχιστο εισόδημα, μιλούμε για λιτότητα, μιλήσανε για λιτότητα. Είναι καιρό σήμερα να ακολουθήσουμε αντίστροφη πορεία και να υπενθυμίσουμε την ισότητα των δικαιωμάτων. Ήρθε η εποχή να πούμε ότι αυτή η οδηγία πλαίσιο είναι σημαντική, διότι δεν υπάρχει εργασία και η εργασία δεν επιτρέπει να βγούμε από την φτώχεια και το ελάχιστο εισόδημα για όλους ε, είναι ένα μέσο κλειδί. Έχουμε λοιπόν εδώ μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσουμε, πρέπει να δράσουμε, διότι σήμερα πρέπει να δράσουμε αποτελεσματικά κατά ε, της φτώχειας και ε, του κοινωνικού αποκλεισμού. Ελπίζω για μια άλλη φορά να μην παρακάμψουμε τις ευθύνες μας. Μερικοί άξονες δράσης κατά τη γνώμη μου πρέπει να έχουν προτεραιότητα. Υιοθετήσαμε σήμερα το πρωί ένα μια προφορικό ερώτημα ε, και μια γνωμοδότηση για τα, στους άστεγους. Αυτή η στρατηγική έχει τη θέση της στην πλατφόρμα και θα μεριμνήσουμε γι' αυτό πέρα από το θέμα των αστέγων ε, που είναι αν θέλετε ο αδύναμος κρίκος ε, ε, για την κατοικία ε, μας δείχνει ότι η πολιτική της κατοικίας, της στέγασης ε, πρέπει να είναι στο επίκεντρο όλων των αποφάσεων και των αποφάσεων των ευρωπαϊκών. Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, εν τέταρτο των Ευρωπαίων θεωρούν ότι μια από τις βασικές αιτίες της φτώχειας ε, είναι η υπερβολική, υπερβολική τιμή των ευπρεπών κατοικιών και 9 στους 10 σκέφτονται ότι η φτώχεια εμποδίζει την πρόσβαση σε ευπρεπή κατοικία η κατοικία αυτή χρειάζεται ε, παρεπόμενες ε, υπηρεσίες για να μπορεί κανείς να ζήσει ευπρεπώς ε, σε μια κατοικία. Πρέπει να έχει καλή τιμή το νερό, ο ηλεκτρισμός, η θέρμανση, οι τηλεπικοινωνίες μεταξύ των άλλων υπηρεσιών κοινή ωφελία πρέπει να είναι εγγυημένε υπηρεσίε και σήμερα πρέπει να αγωνιστούμε για να βρούμε χρηματοδότηση για να καταπολεμήσουμε την επισφάλεια την ενεργειακή. Χρειάζονται ειδικέ απαντήσεις. Πρώτα απ' όλα, η πρόσβαση σε ένα ελάχιστο εισόδημα αυτονομίας επιπλέον. Το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή μας υιοθέτησε ε, την εισήγηση της Εμιλή Τουρίνεν, ε, την αρχή μιας ευρωπαϊκής εγγύησης για την νεολαία, ούτως ώστε να αποφύγουμε η νεολαία η οποία έχει φτάσει και θα φτάσει στην αγορά εργασίας κατά τη διάρκεια της κρίσης, να μην είναι μια χαμένη γενιά. Δεν πρέπει αυτό να παραμείνει ευσεβής πόθος. Οι Ευρωπαίοι πολίτες περιμένουν να περάσουμε από τα λόγια στις πράξεις. Θα ήθελα να αναφέρω ένα από τα μηνύματα κλειδιά του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά της φτώχειας. Ποιος στην ανάλυση του της πρότασης της πλατφόρμας της Κομισιό έλεγε το εξή. Η φτώχεια και ο κοινωνικό αποκλεισμό δεν θα μπορέσουν να μειωθούν με μόνιμο τρόπο, ενώ οι ανισότητε και οι διακρίσει δεν θα έχουν καταπολεμηθεί. Δεν μπορώ παρά να μοιραστώ αυτή την διαπίστωση. Θα πρέπει να μειώσουμε τι διαφορέ τι εισοδηματικέ και του πλούτου και αυτό περνάει από την εξασφάλιση ενός κατάλληλου ελάχιστου εισοδήματος για όλους από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από έναν περιορισμό αυστηρό των υψηλών αμοιβών, τονίζοντας τον περιορισμό των μπόνους. Πρέπει σήμερα να ε, ε, φερθούμε υπεύθυνα ε, και να τονίσουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει αποτρεπτική φορολογία πέρα από ένα κατόφλι θα πρέπει να καταπολεμήσουμε κάθε μορφή διάκρισης στην πρόσβαση στα δικαιώματα, στις υπηρεσίες, στην απασχόληση. Μιλάω για τις κοινότητες που έχουν περιθωριοποιηθεί, για τους μετανάστες. Πρέπει επίσης να εργαστούμε για ένα νέο σκέλος το σκέλος των πολιτικών της πρόληψης. Ποια είναι τα εργαλεία που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για να προλάβουμε αυτή τη φτώχεια. Και τέλος Κλείνω διότι το μέλλον του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Βοήθειας στους Απόρους απειλείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε για το 2012 ένα προϋπολογισμό διαιρεμένο δια του 5 ενώ η ένδια είναι μεγαλύτερη δεν μπορούμε να αφήνουμε, να την αφήσουμε να συνεχίσει ενώ δεν βρίσκεται μια μόνιμη λύση. Εμείς η ομάδα των Πρασίνων θα υποβάλουμε πάρα πολλές τροπολογίες και τελειώνω λέγοντας ότι πρέπει η ανθρώπινη ουσία να μπει στο επίκεντρο των πολιτικών. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, επισύρω την προσοχή σας πάνω στο γεγονός ότι έχουμε να κάνουμε ακόμα με τρεις γνωμοδοτήσεις που πρέπει να συζητήσουμε. Θα σας ζητούσα λοιπόν να είστε πάρα πολύ συνοπτικοί, διότι δυστυχώς ε, δεν θα, μια έκθεση δεν θα παρουσιαστεί. Δίνω τώρα το λόγο. Bye, στην Φρεντερίκ. πάρα πολύ σύντομα, πάρα πολύ θα ήθελα να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η έκθεση. Νομίζω ότι η πρόληψη ε, των αστέγων, ε, η εξασφάλιση κατοικίας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, λόγω της ανεργίας πολλοί χάνουν τα σπίτια τους, λόγω της υψηλής τιμής. Εκτός από τις γενικές υπηρεσίες, επίσης η εκπαίδευση των παιδιών είναι σημαντική, διότι όταν τα παιδιά φτάνουν στο σχολείο καμιά φορά είναι πολύ αργά για να αρχίσουν και, και να μπουν μετά στην αγορά εργασίας. Διακρίσεις, διαχωρισμοί είναι επίσης σημαντικοί και νομίζω ότι θα πρέπει να αναφέρουμε στα εκτιμώντας, όπως αναφέρθηκαν οι Ρωμά, να αναφερθούν αυτά. Αυτό είναι όλο. Ευχαριστώ ε, ε, πολύ. Καλά. Δεν ξέρω ποιος έχει το λόγο τώρα. Εάν ο συνάδελφος Νταρντέν θέλει να κάνει μερικά σχόλια, αλλά σας παρακαλώ να είστε πάρα πολύ σύντομος, ε, θα επανέλθουμε στη συζήτηση Πρόεδρε, θα είμαι πάρα πολύ ε, σύντομος. Θα ήθελα ε, να ευχαριστήσω τους διάφορους παρεμβαίνοντες για τις ιδέες που εξέφρασαν. Έχουμε μια μοναδική ευκαιρία, όπως το είπε η συνάδελφος Ντάλι, και νομίζω ότι θα μπορέσουμε χάρη στις προτάσεις σας και στις τροπολογίες να εμπλουτίσουμε την έκθεση αυτή και χαίρομαι που μπορούμε που θα ξανασυζητήσουμε όλοι μαζί σε μερικές μέρες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Προσθέτω εξάλλου ότι η ημερομηνία, η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι στις 22 Ιουνίου στις 5 το απόγευμα και μετά θα μπορέσουμε να υιοθετήσουμε στην Επιτροπή στις 8 Σεπτεμβρίου αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ σε όλους και τώρα περνάμε στο επόμενο σημείο. Το σημείο 20. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο Συντονισμού της Οικονομικής Πολιτικής. Ο εισηγητής είναι ο πρόεδρο, η πρόεδρός μας στην Οικονομική Επιτροπή Περβάνσιο Σομπέρες επί της ουσίας και ο συντάκτης για γνωμοδότησης είναι ο κύριος Όλε Λούντβιξον που αντικαθίσταται από την κυρία Στάινμπεκ. Σας παρακαλώ ε, με πολύ συντομία να παρουσιάσετε αυτή την εισήγηση. Σας δίνω το λόγο. Ähm, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε ο εισηγητή μα, ο Λε Λούτφιξον, έχει ένα οικογενειακό πρόβλημα και δεν μπορεί να είναι εδώ. Μου ζήτησε όμως ε, να κάνω κάποιε παρατηρήσεις εκ μέρου του. Κατά την άποψή του, θα πρέπει η Κομισιόν να παίξει σημαντικό ρόλο στη διάρκεια αυτού του Ευρωπαϊκού ε, Εξαμήνου. Και εμείς ε, μέσω της γνωμοδότησής μας θα πρέπει να πάρουμε συγκεκριμένη θέση όσον αφορά την, ε, το, ευρωπαϊκό αυτό εξάμεινο στα πλαίσια πάντα και υπό το φως της ε, στρατηγικής 2020. Ε, Πιστεύω ότι θα πρέπει να πάρουμε θέση όσον αφορά την μακροοικονομική κατάσταση και την μικροοικονομική κατάσταση και να δούμε με ποιο τρόπο η οικονομική πολιτική μπορεί να έχει αποτελέσματα στην ε, πραγματική οικονομία. Επίσης, ο κύριος Λούντβικσον θεωρεί ότι στη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θα πρέπει να γίνει σεβαστός ο οικονομικός διάλογος ε, και θα πρέπει οι κοινωνικοί εταίροι να βρουν τη θέση τους, όπως άλλωστε και η συζήτηση την εθνική διάσταση των μισθών και των συντάξεων. Αυτά είναι θέματα τα οποία σαφώς αποτελούν δικαιοδοσία των κρατών μελών. Δεν είναι αποδεκτό, κατά την άποψη του κ. Λούτιξον, άμεσα ή έμεσα ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, απομακρυνθεί από την αρχή της ε, μη επέμβασης σε θέματα που είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Η κοινωνική εταίροι στη διάρκεια της ενσωμάτωσης των οδηγιών θα πρέπει να έχουν δικαίωμα να συζητήσουν ορισμένα ζητήματα Νομίζω ότι το Βέλγιο ήταν η μόνη χώρα ε, η οποία πριν από την μεταφορά των οδηγιών ε, συζητά με τους κοινωνικούς εταίρους και διαβουλεύεται. Είναι η μόνη χώρα. Δεν αρκεί. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο στους σκιώδεις εισηγητές, κυρία Μέρα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Μιλώ εξ ονόματος του συναδέλφου Φιλίπ Μπουλό, ο ε, είναι σκιώδης ε, εισηγητής για το θέμα αυτό του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου Συντονισμού της Οικονομικής Πολιτικής. Ε, στα πλαίσια της εργασίας αυτής λοιπόν για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, ο κύριος ε, Μπουλόν ε, θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρξουν μέτρα για την κατάρτιση και την εκπαίδευση, για την πρόσβαση στην ε, απασχόληση, για την επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας, με τρόπο ώστε από αυτή τη στιγμή πλέον και εφ' να κάνουν σωστές επιλογές τα κράτη όσον αφορά τις βράχοι και μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε σχέση με τα κοινωνικά ζητήματα. Τρεις ε, είναι οι άξονες οι οποίοι παρουσιάζουν ιδιαίτερη σημασία ο άξονας ε, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, ε, κυρίως με καταπολέμηση ή με μέτρα για την καταπολέμηση ε, της αποτυχίας στη διάρκεια του, της σχολικής ζωής και δυνατότητα καλύτερης ένταξης στην αγορά εργασίας μετά το πέρας των σπουδών, εξατομίκευση της διαδικασίας του επαγγελματικού προσανατολισμού. κατάρτιση διαβίου. Πολλής λόγος γίνεται για αυτήν την διαβίου κατάρτιση, αλλά λίγα πράγματα γίνονται επί τόπου. Μέχρι το 2020 θα πρέπει να έχει αλλάξει η κατάσταση και τουλάχιστον να έχει ε, μια καλύτερη ισορροπία η σχέση ζήτησης και προσφοράς. Δεύτερος άξονας, η διευκόλυνση στην πρόσβαση ε, στην απασχόληση και διευκόλυνση όσον αφορά την δημιουργία απασχόλησης. Ε, μέτρα τα οποία θα πρέπει να βοηθούν και εν πάση περιπτώσει να μην εμποδίζουν την ε, δημιουργία απασχόλησης, ε, ένα σύστημα ε, καλύτερης ευελιξίας όσον αφορά την δυνατότητα απολύσεων, έτσι ώστε να παραμείνει σε αρκετά υψηλό επίπεδο η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Επίσης, μέτρα ε, για την ε, καλύτερη ενσωμάτωση των ηλικιωμένων ε, στον, στην αγορά εργασίας, όπως ακριβώς αναφέρεται στις προτάσεις που καταγράφονται στην έκθεση για την ενεργητική γύρανση και βεβαίως συνεχόμενους και διαρκείς διάλογους. Τρίτος σημαντικός άξονας είναι η κοινωνική προστασία με την ιδέα να δημιουργηθεί ένα ελάχιστο ποσοστό κοινωνικής προστασίας που θα ικανοποιεί την, ε, ε, την κοινωνική προστασία των ε, εργαζομένων που βρίσκονται στην χειρότερη θέση και βεβαίως σωστά συστήματα προστασίας από την φτώχεια και προστασία της ποιότητας ζωής. Ο άξονας αυτός είναι πάρα πολύ σημαντικός, ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο της ε, κρίσης ε, που αντιμετωπίζει ε, πλέον η αγορά εργασίας. Θα πρέπει να ενισχυθούν και οι κοινωνικές παροχές αλλά και οι δυνατότητες κοινωνικής αρρωγής προς τους ανέργους κυρίως. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό ήθελα να πει ο συνάδελφός μου. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Μωρέν. Η κυρία Άρκιν παρακαλώ έχει τον λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή που μέσω της συναδέλφου του μας παρουσίασε τις απόψεις, τους, τις απόψεις του. Ναι, βεβαίως ε, χρειαζόμαστε διασύνδεση ε, ανάμεσα στην οικονομική πολιτική, για την κοινωνική πολιτική, για την πολιτική απασχόλησης. Ε, στα διάρκεια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θα πρέπει ο συντονισμός της οικονομικής πολιτικής να έχει καλά αποτελέσματα, να έχει ωφέλη για, τους, για την απασχόληση. Ένα από τα ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζουν πολλές χώρες μεταξύ των οποίων και η δική μου είναι τα μέτρα λιτότητας τα οποία έχουν εφαρμοστεί και βεβαίως ελοχεύει ένας πραγματικός κίνδυνος ε, ε, περαιτέρω από συντονισμού ε, και να παραμεληθούν οι ε, πολιτικές ε, ε, οι οποίες οδηγούν στην αηφορία και την προστασία των κοινωνικών και εκτιμένων. Νομίζω ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να περιληφθούν στα προγράμματα κίνητρα για την δημιουργία θέσεων εργασίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε εργαζόμενους οι οποίοι βεβαίως έχουν την καλή εκπαίδευση, ε, τα σωσ... τις σωστές ε, γνώσεις ε, και αυτή θα είναι η προσφορά και από την άλλη πλευρά να υπάρχουν οι αντίστοιχες θέσεις εργασίας, δηλαδή να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στην προφορά και την ζήτηση. Και άλλα δύο σημεία θα ήθελα να θίξω πιστεύω ότι θα πρέπει να υπογραμμίσουμε τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διάρκεια αυτή της διαδικασία. Είναι το Κοινοβούλιο το οποίο στηρίζει την δημοκρατική ε, λογοδοσία και επομένως θα πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος του Κοινοβουλίου. Αυξάνει το Κοινοβούλιο και την νομιμότητα αλλά και την προσβασιμότητα των ε, ε, πολιτών. Επίσης, εάν δει κανεί τις παραγράφους 1 και 2, υπάρχει κάποια ένταση. Στην 1, ας πούμε, ε, ο εισηγητής λέει ότι θα πρέπει να υπάρξει μια κοινή αντιμετώπιση, των, κοινή προσέγγιση των προκλήσεων. Επίσης, αναφέρεται και στην, στον σεβασμό της αρχής της επικουρικότητας ε, και του κοινωνικού διαλόγου στον τομέα των μισθών και των συντάξεων. Σας λέγω πάντως ότι υπάρχει έτσι μία αμφισημία μεταξύ των δύο. Αυτό που ίσως μπορούμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε στην Επιτροπή μας εδώ είναι να αντιμετωπίσουμε αυτό το σημείο έτσι ώστε να βγει ισορροπημένη η γνωμοδότησή μας. Να έχουμε κοινή προσέγγιση ε, ε, ε, δηλαδή είναι λίγο αμφιλεγόμενο να λέμε κοινή προσέγγιση στη μία παράγραφο και σεβασμό της επικουρικότητας στην άλλη παράγραφο. Είδω. Ναι, μπορούμε να θεωρού, θεωρήσουμε ότι συζητήθηκε το θέμα. Οι τροπολογίες θα παρουσιαστούν μέχρι την 21η Ιουνίου στις 12 ούτως ώστε να μπορέσουμε τον Ιούλιο στην συνεδρίαση της Επιτροπής αυτή τη γνωμοδότηση. Και τώρα περνάμε στο επόμενο σημείο Ε, θα αντιστρέψουμε, θα περάσουμε στο σημείο 22 προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή απασχόληση. Πρόκειται για το σημείο 22 της ημερήσιας διάταξης. Ε, έχουμε ε, το συντάκτη γνωμοδότησης. Όχι. Όχι, τότε <laughs> περνάμε και πάλι στο 21 διότι η κυρία Λίζα Γιακονσάρη είναι μεταξύ μας, προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκών τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεπιχειρησιακής απόσπασης, σημείο 21 και μετά θα ασχοληθούμε με το σημείο που αφορά το συνάδελφο Κοφεράτη. Σας ευχαριστώ. Η οδηγία σας ευχαριστώ. Αυτή η οδηγία εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο του πακέτου μετανάστευσης, είναι αναπόσπαστο τμήμα και είναι καλό η Ευρωπαϊκή Ένωση να θελήσει να έχει μια κοινή πολιτική της μετανάστευσης. Αλλά η προσέγγιση της Επιτροπής είναι πάρα πολύ κατακαιρματισμένη πράγμα που δεν μου φαίνεται ότι είναι καλό. Φοβούμε ότι ε, μια τέτοια προσέγγιση θα μας κάνει να χάσουμε ε, τον μεγάλο προσανατολισμό της οδηγίας, να τον ξεχάσουμε που είναι η προσπάθεια απλούστευσης ε, του όλου συστήματος και η θέσπιση ίσης μεταχείρισης για όλους και φοβούμε ότι πρόκειται να ξεχάσουμε, να παραβλέψουμε αυτό το στόχο και θα ήθελα να το πω στην Επιτροπή. Και εγώ νομίζω ότι είναι σημαντικό να μπορούμε να έχουμε μια κοινή πολιτική της μετανάστευσης, αλλά δεν υποστηρίζω αυτή την προσέγγιση την τομεακή. Νομίζω ότι θα προσθέσουμε νέα προβλήματα αντί να ρυθμίσουμε αυτά τα οποία υπάρχουν. Υπάρχει επίσης το γεγονός ότι εξετάζεται το θέμα ως αν να εξαρτάται από την μετανάστευση. Πράγμα που επηρεάζει την ε, αγορά εργασίας. Είναι δύσκολο να εκτιμηθεί η επίπτωση στην αγορά εργασίας, αλλά πάντως είναι μεγάλη η επίπτωση αυτή. Είναι ο λόγος είναι γιατί το 151 α, β και g πρέπει να προσθεθεί στη νομική βάση εφόσον υπάρχει μια σχέση με την πολιτική της απασχόλησης, πρόκειται για υπηκόους τρίτων χωρών με την Επιτροπή ε, ΛΥΜΠΕ, νομίζω ότι θα πρέπει να προσδιορίσουμε τι εννοούμε με, με στελέχη, εκτελεστικά στελέχη, Για την ώρα οι ορισμοί είναι αμφίσιμοι. Όταν μιλούμε για έναν ζωγράφο, παραδείγματος χάρη, θεωρούμε ότι πρόκειται για έναν εξειδικευμένο εργαζόμενο. Αλλά γιατί χρειαζόμαστε διαφορετικό ορισμό. Η οδηγία για την μπλε κάρτα αναφέρεται α, αναφέρεται σε τέτοιους εξειδικευμένους εργαζόμενους για να δούμε ε, τι είναι το εξειδικευμένο προσωπικό. Υπάρχουν επίσης άλλα θέματα πάνω στα οποία θα πρέπει να επιμείνουμε. σε επίπεδο επαγγελματικό και μετά η αναφορά στην οδηγία περί απόσπασης. Ήμουν Ε, εδώ και 15 χρόνια στην εκπόνηση αυτής της οδηγίας. Ξέρω ότι έθεσε πάρα πολλές δυσκολίες εντωμεταξύ. Η Επιτροπή παρουσίασε μια νέα πρόταση και με τις συνθήκες αυτές ε, μου φαίνεται ότι δεν θα πρέπει ε, να βασιστούμε σε αυτή την οδηγία περί αποσπάσεων. ότι μπορούν να εργαστούν τρία χρόνια στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μην έχουμε μια δεύτερη αγορά εργασίας. Και για να αποφύγουμε επίσης να μην διευκολύνουμε το dumping σχετικά με το δικαίωμα της εργασίας, νομίζω ότι θα πρέπει να πληρώνουμε ε, ίσους μισθούς. Εδώ και μερικά χρόνια ο φτηνότερος μηχανικός στον κόσμο βρισκόταν στην Κίνα. Σήμερα δεν είναι αυτή η περίπτωση. Οι ε, μηχανικοί που κοστίζουν λιγότερο βρίσκονται στην Ουκρανία. Αν έχετε μια γερμανική εταιρεία που θέλει να χρησιμοποιήσει αυτούς τους εργαζόμενους, τους εξειδικευμένους με πολλά προσόντα για να εργαστούν στην Ευρώπη, θα πρέπει θα τους κοστίσει αυτό φθηνότερα να προσλάβουν έναν μηχανικό από την Ουκρανία, από έναν μηχανικό Ούγγρο ή Ισπανικό που είναι ανεργός. Από την ευρωπαϊκή άποψη αυτή δεν είναι μια αποδεκτή προσέγγιση. Δεν χρειάζεται, δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε μια τέτοια κατεύθυνση, διότι η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης είναι αυτό που θέλουμε να βελτιώσουμε εμείς και θέλουμε από τις τρίτες χώρες να μπορούν να προσέρχονται άνθρωποι. Είναι μια καλή αρχή, αλλά δεν μπορεί να οδηγεί σε κάποια στρέβλωση, σε κάποια δηλαδή προτίμηση μόνο φτηνών εργατικών χεριών, φτηνού εργατικού δυναμικού. Αυτές ήταν κάποιες σκέψεις τώρα που εξέθεσα. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο και γι' αυτό δεν προτίθεμαι να μακρηγορήσω και να εξετάσω περαιτέρω λεπτομέρειες. Θα ήθελα μόνο να προσθέσω ότι είναι σημαντική υπόθεση αυτή. Και είναι λοιπόν πολύ σπουδαίο να καταλήξουμε σε μια κοινή ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική. Ταυτόχρονα όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να παρακολύσουμε, να αποφύγουμε να υπάρχει μια διπλοεπικάλυψη ή διπλές, ε, διπλή κανονισμή. Με την επιτροπή λίγο έχουμε καταλήξει σε καλές ε, συμφωνίες για τον, την ίδια δουλειά, ίδιος μισθός και πιο συγκεκριμένοι στόχοι μπορούν να επιτευχθούν με τον συντονισμό αυτό. Στις 21 Ιουνίου καταλήγει η προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών. Ευχαριστώ. Ε, ακριβώς αυτό είναι σωστό όπως είπατε. Αυτή ακριβώς η πρόταση θα μας κάνει να δώσουμε τον λόγο αμέσως στη συνέχεια στο συνάδελφο Κοφεράτη. Έχουμε πάρα πολύ λίγο χρόνο για την παρουσίαση από πλευράς του με πολύ, σύντομο τρόπο τη δική του γνωμοδότηση, που επίσης είναι μια γνωμοδότηση σε σχέση με μια έκθεση της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ για τους όρους όσον αφορά πολίτες τρίτων χωρών για την, την πρόσβαση σε εποχική εργασία στην ε, Ένωση. Ε, ο κύριος Θέρκας. Κύριε Θέρκας, διαδικαστικό κύριος Θέρκας. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο κύριε Θέρκας. Ναι, πρόεδρε. Κατανοώ ότι πιέζει πολύ ο χρόνος σίγουρα και με τη διαδικασία που επισημάνατε πρέπει να είμαστε πολύ σύντομοι. Είναι η μόνη δυνατότητα αυτή για μας. Θέλω να επισημάνω όμως στη γραμματεία ότι την επόμενη φορά που θα έχουμε αυτά τα θέματα στα χαρτοφυλάκια, δύο χαρτοφυλάκια πολύ σημαντικά, θα πρέπει να τεθούν στην αρχή της συνεδρίασης και όχι στο τέλος για να έχουμε κάποιο περισσότερο χρόνο και δυνατότητες να παρέμβουμε και να μην πιέζει ο χρόνος. Ευχαριστώ. Ε, Πρόεδρος, γνωρίζω πολύ καλά ότι αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται, τίθεται με αυτόν τον τρόπο. Έχω εδώ και αρκετούς που ζητούν να παρέμβουν και έχουν εγγραφεί και έχουμε και τον εισηγητή μας ε, από την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, τον κύριο Σαλβατόρε Γιακολίνο και για αυτούς όλους τους λόγους ε, πρέπει να πω ότι έχουμε αυτή τη δυσκολία εδώ να διαχειριστούμε τον ελάχιστο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας καθώς αυτά τα θέματα συνδέονται μεταξύ τους ε, μια και τα δύο αναφέρονται σε όρους ε, και για την ε, πρόσβαση για πολίτες τρίτων χωρών στις εργασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει παρουσιαστεί στο πλαίσιο μιας μεταφοράς και πρόταση οδηγίας σε αυτό το θέμα και στην περίπτωση του κυρίου Κοφεράτη το θέμα είναι για πολίτες τρίτων χωρών για εποχική εργασία μπορούμε να ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση. Απλά όμως ο κύριος Κοφεράτη δεν θα μπορέσει να παρουσιάσει τότε την έκθεσή του. Αυτό είναι το πρόβλημα το οποίο έχουμε. Και γι' αυτό ζήτησα, ζητώ από τον συνάδελφό μας κύριο Κοφεράτη να κάνει την παρουσίασή του και στη συνέχεια θα έδινα τον λόγο στον συνάδελφό μας από την ε, Επιτροπή Λίμπε να παρέμβει και σε όλους τους άλλους ε, που είχαν ε, εγγραφεί μέχρι τις 12.30 γιατί στις 12.30 πρέπει να ολοκληρώσουμε ούτως ή άλλως. Μπορούμε ενδεχόμενα να συνεχίσουμε με τον πίνακα ψηφοφορίας ε, μέχρι τις μία η ώρα, αν θέλετε. Να συνεχίσουμε με αυτή την οδηγία, Πρόεδρε, και μετά με την επόμενη οδηγία για να μην δημιουργηθεί σύγχυση. Δημιουργείται σύγχυση όταν συγχέονται τα πράγματα. Ε, Κύριε Ζήτω συγγνώμη. Πρόκειται για πραγματικά κανθόδη, φλέγοντα θέματα εδώ, που έχουν πολύ μεγάλη σπουδαιότητα και που κινούν τους συναδέφους τους συγκινούν. Δεν ξέρω αν είναι δυνατόν, αλλά αν θα ήταν δυνατόν θα μπορούσαμε μόνο να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση για την πρώτη έκθεση, για το πρώτο θέμα και το απόγευμα στις 3 η ώρα να ξεκινήσουμε το δεύτερο θέμα Εσεί θα αποφασίσετε ποια λίστα θα δώσετε. Εντάξει. Ε, ε, το θέμα είναι της διαχείρισης. Δεν ήξερα αν από τις ε, τρεις θα μπορούσαμε να έχουμε αυτή την δυνατότητα για την αρχή του απογεύματος. Και τώρα θα συνεχίσουμε απλά με την έκθεση που βρίσκεται συζήτηση. Και ευθύς εξ αρχής δίνω τον λόγο λοιπόν για αυτό το θέμα στον κύριο, στον συνάδελφό μας Ευρωβουλευτή της, Ευρωβουλευτή της ΛΥΜΠΕ που είναι συντα... ε, εισηγητής επί της ουσίας. Ζητώ συγγνώμη για αυτό το πρόβλημα χρόνου. Έχετε τον λόγο εσείς παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Άκουσα αυτά όσα είπε η συνάδελφος και εξάλλου έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις, αγαστή συνεργασία Είχαμε μια ακρόαση στις 20 Απριλίου σχετικά με το θέμα αυτό, που με το οποίο ασχολούμεθα τώρα στην Επιτροπή μας και σχετικά με τους εποχιακούς απασχολούμενους που αναβλήθηκε για σήμερα το απόγευμα. Αυτή η οδηγία αναφέρεται στις, ε, στις νόμιμες ε, μεταναστευτικές ροές και στη δυνατότητα πρόσληψης ε, εργαζομένων από τρίτες χώρες που έχουν μια μεγάλη εξειδίκευση που βρίσκουμε δύσκολα στο έδαφος μας. Πιστεύω ότι πρόκειται εδώ για μια οδηγία την οποία θα πρέπει να αναλύσουμε καλά για να κατανοήσουμε τι μπορεί αυτό να μας φέρει. Υπάρχουν ε, τα κρίσιμα σημεία, υπάρχουν ε, ορισμοί οι οποίοι είναι πάρα πολύ γενικοί καμιά φορά, παραδείγματο χάρη η Επιτροπή έχει εκπονήσει κάτι το οποίο είναι καλά ισορροπημένο. Ευχαριστώ την Επιτροπή διότι για τις, τους ορισμούς σχετικά με τους διπλωματούχους, τους ειδικού ε, ίσως ε, θα έπρεπε να παρέμβουμε, αλλά χωρίς να μειώσουμε το πεδίο εφαρμογής, αλλά έχοντας στόχους που να είναι μετρήσιμοι. Αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε στις τροπολογίες που καταθέσαμε το άρθρο 8 για τις ε, ποινές, ε, για τις κυρώσεις. Είναι σημαντικό και υπάρχει και η δυνατότητα εξέτασης ε, των ετοιμάτων του εργαζόμενου που θα ήθελαν να τον συνοδεύσουν ενώ ε, όταν μένει ε, μέχρι τρεις, τρία χρόνια, διότι μπορεί να έχει ένα συμβόλαιο εργασίας, διότι για να έρθει κανείς από την Ινδία, στην Ελλάδα, στην Ιταλία θα μπορούσαμε να έχουμε έξι μήνες. Αντίθετα με τα όσα ήθελε η Επιτροπή που ήταν ένας χρόνος. Θα πρέπει να υπάρχει έξι μήνες χωρίς διακοπή, αδιάλειπτους μήνες. Δεν πρέπει να υπάρχει διακοπή, διότι αυτό είναι σημαντικό και το ξέρουμε αυτό και για την κινητικότητα, αλλά αυτό απαιτεί μια επιπλέον εξέταση και έχουμε το θέμα της κοινοτικής προτίμησης. Πιστεύουμε ότι το κείμενο πρέπει να είναι ενιαίο, απλουστευμένο, βελτιωμένο και είμαστε πεπισμένοι ότι η αμοιβή για δραστηριότητες συγκρίσιμες θα πρέπει να είναι η ίδια διότι δεν είναι αποδεκτό δύο εργαζόμενοι που κάθονται στο ίδιο γραφείο και κάνουν τα ίδια πράγματα να πληρώνονται με διαφορετικό μισθό, διαφορετική αμοιβή. Θεωρούμε λοιπόν ότι η Επιτροπή Αντικτύπου θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβει υπόψη και όλα αυτά τα θετικά στοιχεία της οδηγίας τα οποία βεβαίως ε, ε, πρέπει να συζητηθούν σε σχέση και με τα στοιχεία της οδηγίας ε, για τους εποχικούς εργαζόμενους και βεβαίως τη, όλα τα στοιχεία αυτά λέω να ληφθούν υπόψη. Θα ολοκληρώσω την πολύ σύντομη παρέμβασή μου λέγοντας ότι είναι ουσιώδους σημασίας ε, σε αυτήν την φάση να ληφθούν υπόψη ε, η παρούσα κατάσταση, η ιδιαίτερη κατάσταση όσον αφορά τα αυξημένα μεταναστευτικά κύματα στη Μεσόγειο και επομένως πρέπει οπωσδήποτε να κινηθούμε με ταχύτητα. Επομένως, μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, μαζί με τους σκιώδεις εισηγητές, μαζί με την κυρία Γιά Κονσάρη. Θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει κάτι γρήγορα για Σάρη, θα πρεπει οπωσδηποτε να γινει κατι γρηγορα για αυτους τους εργαζόμενους που αποτελούν πλούτο, που αποτελούν έναν ανθρώπινα έναν ανθρώπινο πόρο πολύ σημαντικό ε, ε, για την, τον οποίο θέλουμε οπωσδήποτε να βοηθήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Σα ευχαριστώ συνάδελφε. Θέλω να σας πληροφορήσω, έχουμε τέσσερις που έχουν ζητήσει να παρέμβουν και έχουν έγγραφει. Ζητώ από κάθε ένα να μην ξεπεράσει τα δύο λεπτά για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτό το σημείο. Μέχρι τις 12.30 ακριβώς. Έχει τον λόγο η κυρία Σρέντερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω για αυτόν τον λόγο αμέσως να ξεκινήσω συζητώντας αυτό το θέμα και να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τις προτάσεις ε, που έκανε. Εργαζόμαστε όμως και στο κείμενο επίσης. Είδα και πάλι πολύ προσεκτικά το, τη διατύπωση του κειμένου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε κάποια ουσιοδέστερα σημεία θα ήθελα να υπησέλθω. Το πρώτο είναι το ότι εγώ πιστεύω ότι αυτό το κείμενο είναι αναγκαίο και με αυτόν τον τρόπο κιόλα, με αυτή τη διατύπωση. Δεν μπορούμε με άλλε διατυπώσει να συγχαίουμε τα θέματα μετανάστευση με τον περιορισμό σε σχέση με τη διαμονή και πολλά κοινωνικά δικαιώματα. Είμαστε πάρα πολύ υπέρ του αυτό το κείμενο θα πρέπει να ισχύει και όχι να αναμειχθεί με άλλα. Δεύτερον, δεν συμμεριζόμαστε την άποψη να αλλάξει οτιδήποτε, διότι ως κοινοβούλιο θα βρεθούμε σε χειρότερη θέση και δεν έχει κανένα νόημα. Η πρόταση είναι δεδομένη. Είναι η ευκαιρία μας τώρα τους κοινωνικούς εταίρους να τους εμπλέξουμε, να συμμετάσχουν. Δεν μπορούμε όλα να τα ξετυλίξουμε και να τα πάμε πίσω στην αρχή. Το τρίτο είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε, σε σχέση με αυτό το κείμενο έκανε κάποια πράγματα που δεν είναι σωστά και μάλιστα καθόλου σωστά. Αυτό το κείμενο δεν πάει ούτε, δεν, δεν είναι καλός, είναι σαφές για ποια ομάδα πρόκειται, ποιες ρυθμίσεις απαιτούνται, αλλά αυτό το κείμενο δεν ανταποκρίνεται σε αυτές τις ανάγκες. Ουσιοδέστατο σημείο και το ανέφερε η συγγήτρια, η οδηγία απόσπασης που έχει αντιγραφεί. Εδώ δεν έχει νόημα αυτό. Πρόκειται για ανθρώπου που εργαζόμενοι έρχονται μέσα στο πλαίσιο της ελευθερίας, της κυκλοφορίας, της διακίνησης και μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι αυτονόητο ότι πρέπει να έχουν τον ίδιο μισθό στον χώρο εργασία τους ε, με άλλους που κάνουν την ίδια δουλειά. Είναι παράλογο να πρέπει να θέλει κανείς άλλα πλαίσια. Δεν ανταποκρίνονται στη λογική αυτής της οδηγίας. Θα αλλάξουμε λοιπόν αυτό το πλαίσιο. Η οδηγία απόσπαση δεν έχει καμιά σχέση με αυτό το θέμα και έτσι θα προσαρμόσουμε εμείς ε, τις ανάγκες στο πραγματικό πλαίσιο. Θέλω να τονίσω ότι θα καταθέσουμε τροπολογίες για το θέμα της κοινωνικής ασφάλειας που είναι το πιο κρίσιμο σημείο, το πιο κέριο σημείο. Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν ισχυρά ασφαλή κοινωνικά συστήματα τα οποία δεν θα διαβρωθούν, δεν θα υπονομευθούν. Τέλος, θέλω να πω κατεπηγόντως ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμείς να έχουμε σωστές μεταφράσεις. Το μόνο κείμενο με το οποίο μπορούμε να δουλέψουμε ως βάση είναι το αγγλικό. Όλα τα άλλα μπορούμε να τα ξεχάσουμε. Είναι τόσο λανθασμένες οι μεταφράσεις που στα γερμανικά υπάρχει και διαφοροποίηση όσον αφορά και την περίοδο παραμονής, Στα αγγλικά είναι τρία χρόνια, στα γερμανικά είναι διαφορετικό το, η χρονική ε, διάρκεια. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει τέτοια διαφορά, τόσο λανθασμένη μετάφραση και είναι τρομερό πρόβλημα αυτό. Ε, θα μπορούσε να κατανοήσει κανείς τα πράγματα όταν του πει κάποιος διάβασε το αγγλικό κείμενο που αποκαθιστά την κατάσταση των πραγμάτων. Όμως είναι κατεπήγον να μπορούμε να δουλεύουμε με σωστά κείμενα, με σωστές μεταφράσεις. Γι' αυτό ζητούμε από την Επιτροπή μας όταν ζητείτε να δουλέψουμε με, με το αγγλικό κείμενο μόνο. Οι άλλε εκδόσεις, οι άλλε μεταφράσεις είναι απόλυτα λανθασμένες. Πρόεδρο, ευχαριστώ. Δίνω αμέσω τον λόγο στον κύριο Κάστλερ αυτό το θέμα για τη μετάφραση είναι ένα πρόβλημα πάρα πολύ σοβαρό και το οποίο τίθεται προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πρέπει πραγματικά να υπογραμμιστεί με κάθε έμφαση όπως έγινε από τη συνάδελφο. Ο κύριος Κάσλερ. Η κυρία Εσαγιά λοιπόν έχει τον λόγο. Παρακαλώ. Από την πλευρά του ΕΛΚΑ ε, ε, θα ήθελα να πω ότι η συντάκτρια Γιακονασάρη έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά ε, και ε, πήρε υπόψη την οδηγία πρέπει να γίνει αυτή η νομοθεσία σε συνεργασία με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και να μελετήσουμε τη λύση αυτή προσεκτικά. Αλλά δεν έχω αμφιβολίες ως προς το θέμα ε, το οποίο ανέφερε στην έκθεσή της ότι θα πρέπει να αφήσουμε ε, τους εποχιακούς εκτός ε, του πεδίου εφαρμογής. Ε, συμφωνώ, οι ορισμοί στο άρθρο 3 θα πρέπει να ληφθούν υπόψη με βάση τις συμφωνίες GATS και να επιτρέπουν μια καλύτερη ταυτοποίηση των κατηγοριών σε αυτές τις μεταφορές. Όπως είπε εδώ ο συγητής, η φράση «uncommon knowledge» Ε, για την προσδιορισμό των ε, ειδικοτήτων ε, δεν είναι νομικός όρος και προσφέρεται για πάρα πολλές διαφορετικές ερμηνείες. Και θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι φράσεις αυτούς τους ορισμούς. Με τον ορισμό στο άρθρο 3 ε, η συγγήτρια Γιάκον Σάρη αναφέρεται ε, σε πάρα πολλά πράγματα και με μερικούς από αυτούς τους ορισμούς συμφωνώ, αλλά θα πρέπει επίσης να έχουμε υπόψη μας ότι αυτές οι δύο οδηγίες ε, έχουν εκπονηθεί για διαφορετικούς λόγους, διαφορετικούς στόχους. Πρέπει να τις μελετήσουμε μαζί για να δούμε αν ε, είναι καλές ε, για αυτόν τον στόχο. Ε, και τελευταίο πράγμα, όχι λιγότερο σημαντικό, διότι δεν έχουμε χρόνο, στο άρθρο 14 η ίση μεταχείριση πρέπει να προσδιοριστεί ούτω ώστε τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης στον χώρο διαμονής να λαμβάνονται υπόψη, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να μην έχει τέτοια πρόβλεψη είχαμε ε, μια παρόμοια συζήτηση ε, για την οδηγία με την ε, ενιαία άδεια και εδώ τα προβλήματα δεν είναι τόσο μεγάλα, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν προβλήματα και τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ναι, και πάντοτε θα πρέπει να θυμόμαστε ότι όλα τα κράτη-μέλη μπορούν πάντοτε να ζητήσουν ευνοϊκότερους όρους για τους εργαζόμενους αυτούς αν το επιθυμούν. Και σε συνεργασία με την, ε, τον εισηγητή, την εισηγήτρια και σκιώδεις εισηγητές ίσως μπορέσουμε να ρυθμίσουμε το θέμα. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ να σέβεστε τα χρονικά όρια. Ο κύριος Κάσλερ και μετά Hirsch. ναι, και από πλευρά μου σχετικά σύντομα. Δύο σημεία θέλω να αναφέρω. Το βρίσκω ουσιαστικά καλό το ότι έχουμε την προσπάθεια που ξεκινά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό τον όρο ότι οι εργοδότες και εργαζόμενοι με την ε, συλλογική αυτονομία για τις συλλογικές συμβάσεις και την αντίστοιχη ελευθερία των ε, συλλογικών εταίρων, συμβατικών εταίρων θα δράσουν. Αυτό είναι η προϋπόθεση. Αυτοδιάθεση των συμβαλωμένων μερών για τις συλλογικές συμβάσεις. Αυτό είναι το αποφασιστικό σημείο. Και σε σχέση με την εισήγηση όσον αφορά την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, όταν ζητούνται κυρώσεις, σταματά η δική μας έγκριση. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε κάτι, πρέπει να υπάρχει σύμφωνη γνώμη των κοινωνικών εταίρων. Δεύτερον, είναι πολύ λόγο και είναι δύσκολο να γίνουν μεταφράσεις και υπάρχουν και λανθασμένες μεταφράσεις ε, και σε αυτά που ανέφερε η κυρία Σουρέτερ και για την χρονική διάρκεια. Θα ήθελα να αναφέρω την έννοια της επιχείρησης. Τι είναι μια επιχείρηση ή και ποια, ποιος είναι ο όρος ε, ε, σε σχέση με τους υψηλά προσοντούχους εργαζόμενους. Αν δεν είμαστε πολύ προσεκτικοί στις διατυπώσεις μας θα υπάρχει σύγχυση και αυτό θα είναι δεδομένο. Πιθανότατα αυτό θα συμβεί. Αυτά ήθελα να αναφέρω. Κατά τα άλλα νομίζω μπορούμε να προσφέρουμε όλοι τη συνεργασία μας ώστε να μην δημιουργηθούν φεεζόνες και να μπορούμε να έχουμε σαφή όρια και για τους εργαζόμενους και για τους εργοδότες. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Τηρήσατε το χρονικό όριο. Η κυρία Ισ, παρακαλώ για να ολοκληρώσουμε. Έχετε τον λόγο. Και εσείς πολύ σύντομα, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και εγώ θα είμαι πολύ σύντομη, μια και ο χρόνος πιέζει τόσο πολύ. Πιστεύω αυτά τα οποία έχουμε μπροστά μας και εγώ όπως και άλλοι χαιρετίζω το ότι έχουμε αυτή την πρόταση τώρα. Θα έλεγα ότι όταν ακριβώς έχουμε θέματα επιχειρήσεων και συζητάμε με τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη και έχουν αρκετές θηγατρικές έδρες στην Ευρώπη αλλά και εκτός Ευρώπης είναι ένα κατεπηγόντος αναγκαίο μέσο ώστε να υπάρξει μια κάποια ελαστικότητα και να μην δημιουργούμε μεγάλη γραφειοκρατική επιβάρυνση που δεν χρειάζεται ώστε κάποιος να αποσπαστεί και να έρθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να κρούσω κόδωνα κινδύνου, να μην είμαστε υπερβολικά διστακτικοί, να μην είμαστε υπερβολικά, στο πω έτσι, για το τι μπορεί όλα να πάνε στραβά. Με την μπλε κάρτα είχαμε στο παρελθόν μια προσπάθεια που ε, οδήγησε σε αυτό το αποτέλεσμα. Είναι μια κατεπίγουσα ανάγκη αυτή για μας να είμαστε αποτελεσματικοί και να δραστηριοποιηθούμε σωστά. Σίγουρα υπάρχουν κάποια σημεία όπου χρειαζόμαστε πιο σαφείς ορισμούς για να δούμε τι μπορεί να γίνει και τι όχι. Σίγουρα και για το τι είναι αναγκαίο. Πρέπει να το ξαναδούμε. Κατά πόσον λοιπόν μπορεί μια οικογένεια να επανενώνεται μέσα στο πλαίσιο αυτών των διατάξεων και κατά πόσον ο ε, συμβίος ή η συμβία θα έχει τέτοια άδεια ή όχι. Αυτά είναι πτυχές που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την ισότητα των γυναικών και την μη διακριτική αρνητική μεταχείριση των γυναικών. Για τις περισσότερες φορές οι γυναίκες συμβίες δηλαδή είναι αυτές που ε, επανενώνονται με την οικογένεια και προσέρχονται στο σύζυγο. Είναι κάποια θέματα τα οποία ούτως ή πρέπει να δούμε, αλλά πιστεύω ότι αυτά μπορούμε να τα κάνουμε μέσα σε ένα πραγματιστικό πλαίσιο προσέγγισης, μέσα στο πλαίσιο της συνολικής παγκοσμιοποίησης και της ανάγκης ανταγωνιστικότητας, να είναι ανταγωνιστική η Ευρωπαϊκή Ένωση και να έχουμε λιγότερους φόβους και δισταγμούς ε, να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Ε, Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι η συνάδελφος, ε, η συγγήτρια παρετείται από την παρέμβαση, δεν θα παρέμβει, σας ευχαριστώ γι' αυτό. Ε, θέλαμε να ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά θα το αφήσουμε για το πλαίσιο της συζήτησης όταν θα έχουμε τις τροπολογίες όταν θα μπορέσουν να παρουσιαστούν, να κατατεθούν μέχρι τις 22 Ιουνίου που είναι η προθεσμία. Ευχαριστώ τους διερμηνείς που μας διευκόλυναν κάποια λεπτά με την παράταση της ε, συνεδρίασης ε, την εργασία μας. Σας ευχαριστώ όλες και όλους και η συνεδρίασή μας θα ξαναρχίσει στις 15.00 στις 3 η ώρα το απόγευμα με την έκθεση του συναδέλφου Κοφεράτη. Σας ευχαριστώ όλους σας. Θα τα πούμε στις 3. Γεια.